Καλησπέρα Ευρώπη. Καλώς ήρθατε στη συζήτηση στη Eurovision. Μένει μόνο μια εβδομάδα πριν από τις ε, εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έτσι σήμερα έχουμε τις μεγάλες ερωτήσεις για αυτούς που θέλουν να ηγηθούν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη πενταετία. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στι Βρυξέλλε, όπου οι έξι υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσουν τι υποψηφιότητέ του. Είμαστε ζωντανή σύνδεση στην Ευρώπη μέσω των μελών τη Eurovision, αλλά μα παρακολουθούν στο ίντερνετ ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Σα καλωσορίζουμε. Είμαστε λοιπόν ε, η Έμιλι Τρανγκουέν από τη French TV. Μάρκους Πράις από τη Γερμανική τηλεόραση και Αναστασίνα Χάικαλα και εργάζομαι στην ανταποκριτριά για την Φιλανδική τηλεόραση στο Παρίσι και θα σα παρουσιάσω τη συζήτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Αλλά βέβαια δεν είναι το θέμα για μα. το θέμα είναι για του υποψηφίου που θέλουν να λάβουν την ε, θέση του επικεφαλής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλωσορίστε λοιπόν τον Νίκο Κουέ Ισπανό που γεννήθηκε στην Ισπανία αλλά είναι Βέλγος ε, συνδικαλιστής από την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Από τη Γερμανία, η Σκά Κέλλερ για τους Ευρωπαίους Πράσινους, δεύτερη φορά στην, ε, στον debate της Eurovision. Από την Τσεχική Δημοκρατία, ο Γιάνν Ζαχράντιλ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμμαχία των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στην Ευρώπη. Από τη Δανία, η Επίτροπος για τον Ανταγωνισμό, Μαργαρέτε Βέσταρ, από την Συμμαχία των Φιλελεύθερων και Δημοκρατικών για την Ευρώπη. Από τη Γερμανία, Μάντφρεντ Βέμπα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επικεφαλής του ψηφοδελτίου του. Και από την Ολλανδία, Φρανς Τίμεμανς, πρώτος αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποψήφιος του κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Αλλά η συζήτηση αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς εσάς παντού στην Ευρώπη. Και εδώ θα ακούσουμε την Αναστίνα. Εγώ θα σα παρουσιάσω λοιπόν τα θέματα για τη μέσα κοινωνική δικτύωση σήμερα το απόγευμα. Είσαστε βασικό τμήμα αυτή τη συζήτηση και για όλο το πρόγραμμα θα παρακολουθώ τα εκατομμύρια Ευρωπαίων που μα παρακολουθούν online, που κάνουν ερωτήσει, που απαντούν και που μα μιλούν μέσα από τον ψηφιακό κόσμο. Πείτε μα λοιπόν τι μετρά για εσά. Χρησιμοποιήστε το hashtag TellEurope για να ακουστεί η δική σα φωνή. Of κάθε debate ε, έχει τους κανόνες του και έτσι και το παρόν. Διαρκεί 90 λεπτά. Ο κάθε υποψήφιος θα έχει από ένα λεπτό για να απαντήσει σε κάθε ερώτηση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, του debate, θα έχει ο καθένας από δύο δυνατότητες να προβάλλουν κάρτα αμφισβήτησης προς δύο υποψηφίους. Και σας παρακαλούμε και εσείς ε, όλοι οι υποψήφοι να αξιοποιήσετε αυτή την ε, κάρτα για να έχουμε μια ζωντανή συζήτηση. Ο καθένας σας θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μια εισαγωγική και μια καταληκτική ομιλία. Και μετά από κλήρωση θα ξεκινήσει ο Νίκο Κουέ από την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Νίκο Κουέ. Είμαι εκπρόσωπος ε, για το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Γεννήθηκα στις ε, Αστουρίες, στη Βόρεια Ισπανία. Ο πατέρας μου ήταν ε, ανθρακορίχος και χρειάστηκε να φύγει από την Ισπανία γιατί ήταν αντίπαλος της ε, φραγκικής δικτατορίας. Και ήρθαμε στο Βέλγιο όπου ε, υπήρξε τρομερή αλληλεγγύη απέναντί μας, Μπορέσαμε να βρούμε ένα χώρο για να σπουδάσουμε, να εργαστούμε και γι' αυτό διαπίστωσα στην πράξη αυτή την αλληλεγγύη που υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτή η Ευρώπη της αλληλεγγύης είναι η Ευρώπη για την οποία αναγωνίστηκα ως ε, συνδικαλιστής. Αυτή η Ευρώπη θέλω να συνεχίσει να υπάρχει. Αλλά δυστυχώς στην Ευρώπη έχουμε επίσης φοροαποφυγή, έχουμε τράπεζες την Ευρώπη των τραπεζών που είναι κατά της αλληλεγγύης. Θέλω λοιπόν μια Ευρώπη που να υπάρχει αλληλεγγύη. Ευχαριστώ Νίκο Κουέ, Ισκά Καλησπέρα σε όλους σας. Αυτό το debate, αυτές οι εκλογές είναι σημαντικές γιατί ο κόσμος από όλη την Ευρώπη κοιτά προς τα μέρος μας και αναζητά λύσεις. Ξέρουν πολλά, ότι πολλά πράγματα πάνε στραβά. Η κλιματική κρίση, η λιτότητα, ε, τα προβλήματα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου. Η Ευρώπη προσπαθεί να ανταποκριθεί στι δεσμεύσει που έχει αναλάβει. Και σήμερα το βράδυ θέλω να σα πω ότι υπάρχει μια διαφορετική Ευρώπη, μια, που, μια Ευρώπη που προστατεύει τον πλανήτη που έχουμε, τον μοναδικό πλανήτη που έχουμε, μια κοινωνική Ευρώπη όπου όλοι έχουν μια αξιοπρεπή στέγαση και αξιοπρεπές εισόδημα. Εμεί, ω πράσινοι λοιπόν μαχόμαστε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου μεγάλε επιχειρήσει πληρώνουν αυτό που του αναλογεί σε φόρο, όπου υπάρχει δικαιοσύνη, όπου υπάρχει σεβασμό και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων. Ξέρω ότι μπορούμε να φτιάξουμε αυτή τη διαφορετική Ευρώπη Ευρώπη, αν τη φτιάξουμε μαζί και μάλιστα με τόλμη. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Γιάννη Ζαχράντη. Καλησπέρα σε όλους. Πιστεύω ότι όλες αυτές τις νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με τα ε, προγράμματα και την ιδέα μια ενωμένη όλο και περισσότερο ενωμένη Ευρώπης που ξεκίνησε ύστερα, ε, πριν από τόσο πολύ, καλό, πολύ καιρό. Έτσι λοιπόν θέλω μια Ευρώπη ευέλικτη, αποκεντρωμένη, μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα σέβεται όλα τη τα μέλη, ανεξαρτήτως το είναι μικρά, μεγάλα, δυτικά, ανατολικά, κράτη-μέλη. Θέλω μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα σέβεται τι εθνικέ κυβερνήσει, η οποία θα συνεργάζεται μαζί του, η οποία δεν θα τις ε, καταπολεμά, δεν θα προσπαθεί να τι ε, η οποία δεν θα προσπαθεί να τους επιβάλλει πράγματα. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα κάνει λιγότερα, αλλά θα τα κάνει καλύτερα, με ε, μια ισορροπία μεταξύ του εθνικού και του ευρωπαϊκού επίπεδου. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία είμαι διατεθειμένος, έτοιμο και ικανός να εξασφαλίσω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάργαρετ Βεστάγερ. Είμαι η Μαργαρίτα Φερστέγκα από τη Δανία Έχω μαζί με τον σύζυγό μου τρει κόρε. Ήμουν υπουργό, πολιτικός ηγέτη. και σήμερα εργάζομαι για εσά ω επίτροπο Ανταγωνισμού. Εξασφαλίζω ότι ακολουθούν του κανόνε οι επιχειρήσει. Εσεί, ω καταναλωτέ, λοιπόν έχετε την επιλογή, έχετε την ποιότητα και τι δίκαιε τιμέ. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να έχετε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ζείτε τη ζωή που θέλετε στην κοινότητά σας, να αισθάνεστε ότι έχετε το δικαίωμα αυτό. Η Ευρώπη είναι το καλύτερο μέρο για να ζει ε, σήμερα, ιδιαίτερα ω γυναίκα. Έχουμε πετύχει πραγματικά τόσο πολλά. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι όλα πάνε καλά. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματο, το θέμα τη τεχνολογία, να δημιουργηθούν κοινωνίε βάσει κράτου δικαίου, όπου θα μπορούμε να προβλέπουμε για εσά ό,τι χρειάζεστε στην καθημερινή σα ζωή. Γι' αυτό είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο Manfred Βέιμπα. Σας ευχαριστώ. Το τελευταίο διάστημα πήγα σε πολλές χώρες της Ένωσης και συναντήθηκα με πολλούς Ευρωπαίους. Και διαπίστωσα ότι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες, τους ίδιους φόβους, αλλά και τις ίδιες ελπίδες για το μέλλον της Υπήρου μας. Και αυτό που εννοώ είναι να σας εξηγήσω με τι μέθοδο θα αντιμετωπίσω το θέμα αυτό. Θέλω η Ευρώπη να είναι κοντά στους πολίτες, να ενδιαφέρεται για τα καθημερινά θέματα των πολιτών. Μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή των συμπολιτών μας. Αυτό θέλω. Και νομίζω ότι ο τωρινός πρόεδρος της Κομισιόν, ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, αποκάλεσε την Ευρωπαϊκή του Επιτροπή Επιτροπή της τελευταίας ευκαιρίας. Είναι από τη δική μας ε, πολιτική οικογένεια. Εγώ θέλω η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας νέας απαρχής όπου θα έχουμε αισιοδοξία. Θέλουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε πολλά ως Ευρωπαίοι. Ευχαριστώ Μάνφρετ Βέμπερ και εν τέλει ο Φραν Τίμερμανς. Χαίρετε και καλησπέρα. Ξέρετε, στην παλάμη του χεριού σας κρατάτε την Ευρώπη, το μέλλον της Ευρώπης. Την επόμενη εβδομάδα θα ορίσετε το μέλλον της Ευρώπης για την επόμενη πενταετία. Για εκείνους που λένε ότι η Ευρώπη και οι περιβολίτες της είναι καλύτερο να, έχουν, να μην έχουν Ευρωπαϊκή Ένωση, του συμφέρει δηλαδή να καταρρεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν άδικο. Ούτε πιστεύω ότι χρειάζεται να αλλάξουμε ιδέες. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή, μια ισχυρή Ευρώπη με θεμελιώδη μεταρρύθμιση της Ευρώπης. Ήρθε πια η ώρα να αρχίσουν να πληρώνουν πληρώνουν φόρο οι επιχειρήσεις. Ήρθε πια η ώρα να εισηχθεί ένας ελάχιστος μισθός σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχει έρθει πια η ώρα να εξασφαλιστεί ισότιμη αμοιβή για άνδρες και γυναίκες, να καταπολεμηθεί η βία κατά των γυναικών. Ήρθε πια η ώρα να ενισχυθεί το κράτος δικαίου σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ισχύουν οι νόμοι για όλους. Ήρθε πια η ώρα το κλίμα, η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον να μπουν στο επίκεντρο των μελημάτων της προσεχούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό έχω να σας προτείνω για απόψε. Ευχαριστούμε. Φραν και σας ευχαριστώ όλους για τις τοποθετήσεις σας. Η συζήτηση αυτή λοιπόν το debate γίνεται και για σας και μέσω ημών με το διαδίκτυο. Παρακαλώ λοιπόν την Αναστήνα να αναλάβει τώρα να μας δώσει κάποιες αντιδράσεις, κάποια πρώτα tweets για τη συζήτηση. Ναι, Εμίλη, και καλώ ορίσατε στον κόμβο μέσω κοινωνική δικτύωση. Όπω βλέπετε, παρακολουθούμε όλα τα σχόλιά σα, όλε τι ερωτήσει σα, ε, εγώ και η ομάδα μου. Και ναι, όντω η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι πάρα πολύ ζωντανή. Έχουμε πολλέ ερωτήσει. Ε. Έχουμε λάβει ήδη πολλέ ερωτήσει και πριν ξεκινήσει καν το debate ε, στο hashtag Tell Europe το οποίο ήδη είναι σε κορυφαίο επίπεδο στη Γερμανία και στο Βέλγιο και φαντάζεστε, όπως φαντάζεστε έχουμε κάποια θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή online. Δεν ξέρω αν φαντάζεστε ποια είναι. Να σας πω, το Brexit. Αλλαγή κλίματος, η σφαίρα ιδιωτική στο ψηφιακό κόσμο και η μετανάστευση. Και η Sea-Watch έχουμε στο hashtag Europe ότι έχουμε ε, σώσει σήμερα 65 άτομα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί προφανώ μεγάλο ζήτημα. Να ακούσουμε λοιπόν και τη δική σα φωνή. Να χρησιμοποιήσετε λοιπόν το hashtag Tell και α επανέλθουμε στο debate. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ Αναστίνα για αυτή την πρώτη ματιά στο τοπίο των κοινωνικών μέσων. Και τώρα θα περάσουμε στην μετανάστευση, που είναι το θέμα που ανέφεραν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι στι δημοσκοπήσεις για τι ανησυχίε του. Αλλά η Ευρώπη δεν μπόρεσε να βρει μια κοινή πολιτική λύση. Η ιδέα της επανεκατάστασης ε, αντιμετωπίζεται με αντίσταση και ακόμη για μερικές δεκάδες ε, μεταναστών που φτάνουν με καράβια όπως το Aquarius ή του Sea Watch βλέπω ότι οι κυβερνήσεις δεν θέλουν να τις πάρουν. Οπότε η ερώτησή μου, επειδή υπάρχουν αυτές οι εντάσεις για τη μετανάστευση, εσείς ως πρόεδροι της Επιτροπής θα σταματούσατε τις προσπάθειες να υπάρξει κοινή λύση και αν όχι πώς θα λύσετε το πρόβλημα και να απαντήσει πρώτος ο κύριος Ζαχράντιλ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι δεν θα επαναλάβω τα ασφάλματα της ε, τρέχουσας Επιτροπής με την εισαγωγή υποχρεωτικών ποσοστώσεων υποδοχής μεταναστών που δυστυχώς δεν έφεραν αποτέλεσμα και δυστυχώς ακόμη ε, ενίσχυσαν τους διχασμούς στις διαιρέσεις μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση που θα κάνει σεβαστά τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών και των εθνικών κοινοβουλίων να αποφασίζουν αν θέλουν να χορηγήσουν ή όχι το άσυλο, την προσωρινή ή τη μόνιμη δυνατότητα εγκατάστασης ή ακόμη και την ηθαγένεια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όμως είναι να καταπολεμήσουμε πάνω απ' όλα την διακίνηση μεταναστών, το εμπόριο ανθρώπων, να ανοίξουμε κέντρα υποδοχής ε, εκτός Ευρώπης, ιδάλλως δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την ε, λαθροδιακίνηση και το εμπόριο ανθρώπων. Πρέπει να βρούμε λύσεις με συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες χώρες που θα το δεχθούν. Πρέπει να συνεργαστούμε στενά μαζί τους και πάνω απ' όλα πρέπει να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση στην Αφρική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαχράντιλ. Κύριε Βέμπερ, εσείς τι θα κάνετε. Η μοναδική ευκαιρία είναι μια ευρωπαϊκή λύση, γιατί δεν χωράει η αφιβολία. Και έχουμε δύο βασικού πυλώνε στο Ευρωπαϊκό Λογικό Κόμμα. Ο πρώτο πυλώνα είναι να ε, υπάρχει άφηξη και έλεγχο τη άφηξη των μεταναστών από τα κράτη. Γι' αυτό ζητήσαμε λοιπόν 20.000, 10.000 υπαλλήλου τη Frontex. Το δεύτερο θέμα είναι τι γίνεται στη Μεσόγειο, στη Λαμπεντούσα. Αυτό που μα ε, υπενθυμίζει ποια είναι η ευθύνη μα σε ό,τι αφορά την τον ανθρωπισμό θα πρέπει να λάβουμε τι ευθύνε μα αυτέ. Αυτό σημαίνει ένα μεγάλο σχέδιο Marshall για την Αφρική. Θέλω έναν επίτροπο, ο οποίο θα έχει κατά νου μόνο τα αφρικανικά συμφέροντα, για να ξεκαθαρίζει και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουμε αυτό ω προτεραιότητα. Έχουμε λοιπόν την έλεγχο των συνόρων και την ανθρωπιστική αντίδραση. Και η Άγγελα Μέρκελ, καγκελάριο τη Γερμανία, έδειξε ότι αναλαμβάνουμε τι ευθύνε μα. Και μαζί με τον Ζαν Κλοντ η Άγγελα Μέρκελ κατέδειξε ότι είμαστε έτοιμοι να έχουμε και συμφωνία με την Τουρκία για να ελέγξουμε το τι γίνεται στα σύνορά μα. Και τα αντίστοιχα στοιχεία λοιπόν αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ. Κύριε Κουέ, εσεί θα σταματούσατε τι προσπάθειε για κοινή λύση. Ε, Υπενθυμίζω ότι η μετανάστευση είναι πρώτα απ' όλα ένα τρομερό ανθρώπινο δράμα. Και εγώ είμαι πατέρα παράνομου μετανάστη, γιατί ήρθε χωρί χαρτιά ο πατέρα μου στην. Συγγνώμη, γιο παράνομου μετανάστη, γιατί ο πατέρα μου ήρθε χωρί χαρτιά. Ακόμη και χθε ε, βυθίστηκε ένα καράβι και 50 άτομα έχασαν τη ζωή του. 30.000 έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο. Η ευρωπαϊκή ευθύνη είναι πολύ σημαντική. Όλε οι πολιτικέ που οδήγησαν στην αποσταθεροποίηση τη γειτονία μα πρέπει να επανεξεταστούν για την Ευρωπαϊκή Αριστερά θεωρούμε ότι η μετανάστευση είναι μια δυνατότητα, μια ευκαιρία. Είμαι εγώ ένα παράδειγμα. Είναι μια δυνατότητα για πολλούς που δεν έχουν τη δυνατότητα στη χώρα προέλευσής τους να αναπτυχθούν. Για μας δεν τίθεται θέμα εισβολή στην Ευρώπη. 0,5% του πληθυσμού μας είναι μετανάστες και μπορούν να συμβάλλουν στην ανανέωση της Ευρώπης. Για μας και για μένα που είμαι γιος μετανάστη θεωρώ ότι η δηλώσει του κυρίου Βέμπερ που είναι υποτίθεται μια τελική λύση είναι αρκετά απαράδεκτες. Ευχαριστώ κύριε Κιουέ. Κύριε Βεστάγιαρ. Τι θα κάνετε για αυτούς που κάποτε μπήκαν σε ένα καράβι για να φτάσουν όπως ε, οι γονείς του κύριου, ε, του Κουέ. Κύριε Βεστάγιαρ νομίζω ότι το σημαντικό είναι να βρούμε τι λύσει τι μακροπρόθεσμες και να τι αντιμετωπίσουμε με την ίδια αίσθηση επίγοντος όπω η διάσωση στη θάλασσα. Η θάλασσα δεν πρόκειται ποτέ να δοθεί λύση. Η μετανάστευση θα υπάρχει για πάντα λόγω τη κλιματική αλλαγή, λόγω των αλλαγών στι οικονομικέ συνθήκε. επίσης. Το πιο σημαντικό όμω. και βλέπω ότι οι Ευρωπαίοι έχουν μια μεγάλη καρδιά, καρδιά ανοιχτή για τους πρόσφυγες, να δώσουν προστασία δηλαδή σε αυτούς που τη χρειάζονται και ταυτόχρονα όμως περιμένουν από εμά να βρούμε τρόπους να διαχειριστούμε τη μετανάστευση και να δώσουμε νόμιμες λύσεις για τη μετανάστευση. Δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους που μπαίνουν και βγαίνουν στην Ευρώπη χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι ή πώς. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κοινέ λύσει, ένα κοινό σύστημα ασύλου, κοινή αλληλεγγύη. Μπορούμε να συζητήσουμε το πώ θα το εξασφαλίσουμε αυτό. Αλλά από κοινού οφείλουμε να το πράξουμε, ιδάλω θα αποτύχουμε. Ευχαριστώ, Μαργέτε. Ακούσαμε πολλά για το τι θα έπρεπε να κάνουμε. Φρανς Τίμερμανς, που είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φρανς Τίμερμανς, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα αν ήσασταν εσείς πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά την κάθε φορά που κάθε ένα άνθρωπο στην ε, Μεσόγειο, η Ευρώπη χάνει ένα κομμάτι τη ψυχή τη. Χάνουμε τι αξίε μα. Κατά δεύτερον, όταν ο κόσμο βρεθεί σε ένα καράβι στη Μεσόγειο, αναγκαστικά θα πρέπει να του φροντίσουμε του ανθρώπου αυτού. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πρόστιμα σε ψαράδε και άλλε βάρκε που σώζουν ζωέ, όπω γίνεται στην Ιταλική κυβέρνηση. Είναι απαράδεκτο αυτό. Κατά τρίτον, θα πρέπει να αποτρέψουμε ο κόσμο αυτό να μπαίνει καν στα καράβια αυτά. Και γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Μαύρετ Βέμπερ συμφωνώ μάλλον μαζί του, ότι χρειαζόμαστε ένα σχέδιο για την Αφρική. Αυτό έχει να κάνει με τη μοίρα τη Ευρώπη. Αλλά και η καλύτερη φυλακή και όλε οι συμφωνίε του κόσμου δεν θα μα βοηθήσουν. Χρειαζόμαστε και αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Η αλληλεγγύη όχι μόνο για πράγματα που μα αρέσουν. Η αλληλεγγύη, ξέρετε, είναι και για πράγματα που δεν μα αρέσουν. Και οι κεντρικέ, μάλλον αν συνεχίσουν κάποιε χώρε τη κεντρική Ευρώπη να αρνούνται την αλληλεγγύη, ε, αργά ή γρήγορα θα έχουμε πάλι σύνορα στην Ευρώπη, εκεί που δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Και αυτό θα είναι προ ει όλων των πολιτών Χρειαζόμαστε λοιπόν να το αποτρέψουμε αυτό και χρειαζόμαστε αλληλεγγύη. Thank you. Thank you, Ευχαριστώ πολύ, Φραντ Τίμερμαντς. Η Σκά Κέλλερ. Εσείς, ως πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα κάνατε. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και πρέπει να υπάρχει δίκη κατανομή των ευθυνών. Και πρέπει να στηρίξουμε και τις τοπικές κοινωνίες που κάνουν τόσο πολλά για να υποδεχθούν τους μετανάστες ε, πολλές ε, τοπικές κοινωνίες κάνουν πολλά αυτό που είναι απόλυτα παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει τώρα στη Μεσόγειο όπου πνίγονται άνθρωποι και ξέρουμε που είναι καλούν το κέντρο έρευνα και διάσωση και κανεί δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Οι Ιταλοί του λένε να τηλεφωνήσουν στη Λιβύη και στη Λιβύη δεν απαντάει κανεί. Γιατί υπάρχει εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη, δεν υπάρχει ακτοφυλακή. Και σε αυτέ τι πολιτοφυλακέ που αποκαλούνται ακτοφυλακή, δίνουμε στήριξη. Πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή προσπάθεια έρευνα και διάσωση. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε ούτε ένα άτομο να πνίγεται στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ, Σκακέλερ. Ευχαριστώ για τον πρώτο γύρο των απαντήσεων. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με την ανεργία των νέων. Αν κοιτάξουμε στη λεπτομέρεια, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό, μια τεράστια διαφορά μεταξύ των κρατών του Βορρά και τη Ανατολή. Όπω η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία, ακόμα και η Γαλλία, η ανεργία των νέων, παραδείγματι στην Ελλάδα, έχει φτάσει στο 39%. Τι εξαγήσει όμω μπορεί να δοθεί σε αυτό είναι ήταν υπερβολική λιτότητα όπως στην Ελλάδα ή την Πορτογαλία ή μήπως δεν έγιναν αρκετές μεταρρυθμίσεις όπως ίσως συνέβη στη Γαλλία και την Ιταλία. Ερώτηση λοιπόν προς τους υποψηφίους πώς θα προσπαθήσετε να εξασφαλίσετε και πάλι θέση εργασίας για τους περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια νέους Ευρωπαίους. Κύριε Ζαχάντη, έχετε το λόγο. Καταρχάς, να πω ξεκάθαρα ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό προς την επιχειρήση με καλή νομοθεσία, με καλά προγράμματα από τον προπολογισμό. Κάποια προγράμματα είναι ήδη, έχουν ήδη αναπτυχθεί. Έχουμε την ψηφιακή Ευρώπη, Digital Europe, 10 δις ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε επίσης τον ορίζοντα Ευρώπη που υποστηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη με άλλο τμήμα του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Και έχουμε επίση και το InvestEU, επενδύσει στην Ευρώπη, που ε, συνδυάζει δημόσιου και ιδιωτικού ε, πόρου για την βελτίωση των υποδομών. Πιστεύουμε, πιστεύω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε εξειδικευμένε λύσει για κάθε χώρα, γιατί οι οικονομίε μα είναι πολύ διαφορετικέ. Είναι διαφορετικέ οι δομέ τη οικονομίας λοιπόν και κοιτώντα τι γίνεται στην Ευρώπη βλέπουμε ότι σε κάποιε χώρε ε, υπάρχει περιβαλλοντικό δίκαιο κάτω από 3% στη χώρα μου. Άρα εξειδικευμένε λύσει. Ε, και καλή νομοθεσία, καλά προγράμματα. αυτέ είναι οι λύσει που έχω να προσφέρω. Ευχαριστώ Γιάνν Ζάχναντιλ. Και τώρα ο Μάχρετ Βέμπερ από τη Γερμανία. Η Γερμανία πάντα επιμένει ε, ότι πρέπει να τηρείται το κριτήριο του 3% επιμένει στη λιτότητα. Δεν προκαλεί αυτό την ανεργία στον Νότο. Θα αλλάξετε κάτι. Πρέπει να θυμίσω ότι οι Γερμανοί, οι Δανείοι, οι Αυστριακοί και οι Φιλανδοί τα πάνε πολύ καλά οικονομικά. Ένα καλό μέλλον υπάρχει μόνο αν υπάρχει ανάπτυξη, ιδιαίτερα για τους νέους. Από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Χρειάζεται και ευθύνη και αλληλεγγύη. Από κοινού θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ένα θέμα, για παράδειγμα, που είδα στο Πόρτο, στην Πορτογαλία. Συναντήθηκα με φοιτητέ και μου είπαν ότι Φραντς το κύριο για αυτούς δεν είναι ελάχιστο μισθός, όπως λένε οι σοσιαλιστές. Θέλουν καλούς μισθούς και θέσεις εργασίας για να μπορέσουν να φτιάξουν οικογένειες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε σωστή οικονομική πολιτική που να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει υποδομές, σημαίνει έρευνα, σημαίνει ανοιχτό εμπόριο. Χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή ενιαία αγορά για το μέλλον. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ, Μάνφρετ Βέμπερ, και σα υπενθυμίζω ότι έχετε δύο κάρτε ένσταση ε, για του ε, συνομιλητέ σα, συνυποψηφίου σα. Νίκο Κουέ, συμφωνείτε με τον ε, Μάνφρετ Βέμπερ, μια καλή οικονομική πολιτική αρκεί για να εξασφαλιστεί η απασχόληση στην Ευρώπη. Απάντηση. Όχι, δεν νομίζω. Είναι πολύ καιρό τώρα που το κόμμα του έχει την εξουσία στην Ευρώπη και δυστυχώ οι πολιτικέ αυτέ δεν είναι αποτελεσματικέ. Βεβαίω γίνονται ωραίε ομιλίε κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά μετά επανέρχεται η λιτότητα, η μεταρρύθμιση τη αγορά-εργασία, των ε, συνθήκων επισφαλού απασχόληση με μισθού που είναι χαμηλότεροι και από τον κατώτατο μισθό και αυξάνεται και η ηλικία για τη σταξιοδότηση για τους γονείς που θα μείνουν να δουλεύουν μέχρι τα 65 έτη ηλικίας ενώ οι νέοι, τα παιδιά τους δηλαδή, είναι άνεργοι και μένουν στο σπίτι. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτή η αβεβαιότητα, η επισφαλή συνθήκες εργασίας πρέπει να σταματήσουν οι συμβάσεις μηδενικών ορών που δεν οδηγούν πουθενά, να βρούμε πραγματικές θέσεις εργασίας, να υπάρχει ένας πραγματικός κατώτατος ευρωπαϊκός μισθός πάνω από το όριο τη φτώχεια. Ιδάλω, αν είναι να συνεχίζει κανεί να εργάζεται για να μένει πάντα φτωχό, θα ήταν παράδεκτο για όλου αυτού του νέου. Και πρέπει αυτέ οι συμβάσει αόριστου χρόνου εργασία να είναι ο πραγματικό στόχο για όλου αυτού του νέου στην Ευρώπη. Ευχαριστώ που, πολύ, Νίκο Κουέ. Μαργρέτε Φέσταγκερ, μέσω του γενικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος μπορούμε να δώσουμε απάντηση στα εκατομμύρια νέων Νομίζω ότι και τα δύο μπορούμε να τα πατήχουμε, γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ενωθεί για να εξασφαλίσουν ότι σε κάθε χώρα θα υπάρχει προσφορά εκπαίδευσης, κατάρτισης και συγκεκριμένων θέσεων απασχόλησης. Γιατί δίχως ε, θέσεις ε, απασχόλησης δεν υπάρχει και μέλλον. Και φυσικά είναι πολύ εύστοχο ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή οικονομία. Πρέπει να επενδύσουμε για να υπάρχει περιθώριο ανάπτυξη για τι επιχειρήσει και βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, νέε θέσει απασχόληση, 12 εκατομμύρια νέε θέσει απασχόληση στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αλλά πολλέ από αυτέ δεν είναι καλαπληρωμένε. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια οικονομία όπου κανεί να μπορεί να βγάζει ένα καλό εισόδημα, ξεπρεπέ εισόδημα όταν δουλεύει ε, σε καθεστώ πλήρου απασχόληση. Και εδώ έρχεται η συζήτηση για το κατώτατο μισθό. Έχουμε διαφορετικά συστήματα. Είναι σημαντικό να το σεβαστούμε αυτό, γιατί θα πρέπει να καλέσουμε του κοινωνικού εταίρου να μα βοηθήσουν, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε αυτή μπορεί να πετύχει κάτι, αλλά μόνο μαζί με τα κράτη-μέλη μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Thank you, Margaret Ευχαριστώ, Margaret Φεστάγκερ. Φραν Timmermans. παρακαλώ, ω αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ω ενδεχόμενα μελλοντικό πρόεδρο, μπορείτε να απαντήσετε. Όταν πήγα στην Πορτογαλία, οι νέοι με ρωτούν ότι όταν ο Αντώνιο Κώστα θέλει να δημιουργήσει περισσότερη ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη και του είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίω να το κάνει. Ενώ ο Μάφρετ δεν είπε όχι, να τιμωρηθεί η Πορτογαλία. Αλλά επανέρχομαι για τους νέους. Πολύ συγκεκριμένα. Το έρασμος πρέπει να επεκταθεί για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από το εάν είναι μαθητές, φοιτητές, αν έχουν δουλειά ή όχι. Έτσι θα μπορέσουν να μάθουν από άλλε χώρε. Και πρέπει να υπάρχει ελάχιστο μισθό που να είναι στο 60% του μέσου μισθού. Αυτό θα προστατεύσει του νέου από δουλειέ που πληρώνουν 2-3 ευρώ την ώρα. Επίση, να επεκταθεί το πρόγραμμα εγγυήσεων για την απασχόληση των νέων. Έχει επιτύχει πολλά. Πρέπει να επεκταθεί και να μειωθεί στα 16 η ηλικία ψήφου για να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο στις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Ευχαριστώ πολύ, Φρανς Τίμερμανς. Μα νόμιζα ότι συμφωνούσαν σε όλα, αλλά όχι. Είδαμε ότι ο Βέμπερ έκανε ήδη ένσταση. 30 δευτερόλεπτα Μάνφρετ και μετά 30 δευτερόλεπτα του Φρανς Τίμερμανς. Μάλιστα, μας λέτε δηλαδή ότι η αλληλεγγύη είναι η λύση για την Ευρώπη, αλλά δεν μιλάτε για υπευθυνότητα. Θα, υπενθυμίσω όμως ότι ο Επίτροπο ο αρμόδιο για τα θέματα αυτά και ο Ντάισελμπλουμ, ο οποίο είναι πρώην συνάδελφος του Τίμερμαν, όταν ήταν πρωθυπουργό των κατοχωρών, επικεφαλή του Eurogroup, ήταν αυτοί οι οποίοι ανέλαβαν τι ε, δύσκολε αποφάσει και ο πρωθυπουργό τη Πορτογαλίας, Σοσιαλιστή και πάλι πρώην πρωθυπουργό, είναι αυτό ο οποίο είναι επικεφαλή τώρα του Eurogroup του σώματο που είναι υπεύθυνο για να αναλυφθούν τα απαραίτητα βήματα. Πρέπει ο καθένα λοιπόν να αναλάβει τι ευθύνε του και οι σοσιαλιστέ να υλοποιούν τις πραγματικέ τους πολιτικές. Κύριε Τίμερμαν, μπορείτε να απαντήσετε. Μα δεν έχει καμία σχέση με αυτά που είπα. Ο Πιέχ Μασκοβισή κοίταξε τα σχέδια. Είπε ναι, μια χαρά. Ο Ζαν Κλοντ Ιουνκέρ είπε το ίδιο για τα σχέδια για την Πορτογαλία. Αλλά ο Μάνφρεντ Βέμπερ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα απέρριψε. Είπε όχι, πρέπει να τιμωρηθεί η Πορτογαλία, να μην γίνει αυτό που προτείνει η Επιτροπή. Αυτό συνέβη. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι πολύ μεγαλύτερη τώρα και έχουν αυξηθεί και οι θέσει εργασία στην Πορτογαλία γιατί εγκατέλειψαν τη λιτότητα και αυτό πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσει. Ευχαριστώ πολύ. Φρανς Τίμερμανς και τελευταία επ' αυτών η Σκάκελε. Παρακαλώ. Νομίζω ότι τα μέτρα λιτότητα τα οποία ελήφθησαν στην Ευρώπη πραγματικά έκαναν μεγάλη ζημιά. Έκαναν μεγάλη ζημιά στον κόσμο προσωπικά. Έχασαν τη δουλειά τους νέοι άνθρωποι, όχι όμω μόνο νέοι άνθρωποι. Ήταν ένα μεγάλο πλήγμα όμως και στην ε, ευρωπαϊκή αυτή, ε, στο ευρωπαϊκό όνειρο για την ε, κοινή ευημερία. Να μην ξεχνάμε λοιπόν, αν, νέοι, αν οι νέοι είναι άνεργοι, αυτό σημαίνει ότι θα έχουν χαμηλότερο εισόδημα και στο μέλλον. Άρα η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων είναι ένα βασικό θέμα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο για κάποιες περιφέρειες και για κάποια κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η εγγύηση για τους νέους να είναι δεσμευτική για όλου να έχει σωστή χρηματοδότηση και να πρέπει να, έχουμε, να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τι σωστέ δουλειέ στο μέλλον, να επενδύσουμε στην πράσινη οικονομία. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα δημιουργηθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Γιατί να περιμένουμε λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε τέτοιε επενδύσεις οι οποίε πραγματικά θα έχουν ως στόχο την κοινωνική και οικονομική μετάβαση τη οικονομία μα. Ευχαριστώ Γιάννη Ζαχράντιλ. Θέλετε να πείτε κάτι με την κάρτα. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Τίμερμανς. Συμφωνείτε ότι ποικίλει ιδιαίτερα από κράτος μέλος σε κράτος μέλος η ανεργία. Σε άλλες χώρες είναι πάνω από 10% και άλλες χώρες είναι στο 3%. Θεωρείτε ότι αυτό αποδεικνύει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά ε, κοινοβούλια είναι σε καλύτερη θέση να βρουν τις πιο προσαρμοσμένες λύσεις για την αγορά εργασίας τους από ό,τι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ναι, αν είχαμε εφαρμόσει την ίδια λογική για τα διευθυντικά ταμεία για τα κράτη-μέλη πριν από 15 χρόνια, τότε η τσεχική δημοκρατία δεν θα ήταν τόσο ευημερούσα όσο είναι τώρα και η ανεργία σα δεν θα ήταν τόσο χαμηλή όσο είναι. Χωρί τα διευθυντικά ταμεία θα είχατε επιτύχει αυτό που επιτύχατε. Αυτό ακριβώ είναι έκφραση τη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν συμφωνείτε ότι είναι επίση έκφραση τη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη όχι να λέμε έχουμε χαμηλή ανεργία, αλλά μας ενδιαφέρει και το γεγονός ότι στην Νότια Ευρώπη είναι πολύ ψηλή η ανεργία, 30% των νέων και θα βοηθήσουμε και αυτούς. Ευχαριστώ πολύ Φραν Τίμερμανς και ελπίζω να καταλαβαίνετε γιατί σας ενθαρρύνω να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες ένσταση για να γίνει ουσιώδη συζήτηση. Σα ευχαριστώ όλου, ευχαριστώ Σκακέλερ, σας ευχαριστώ όλου για τι πρώτε απαντήσει για τη μετανάστευση και για την ανεργία των νέων. Τώρα ε, περνάμε από τη συμβατική αντιμετώπιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πραγματικά πολύ ε, έντονη η αντίδραση όλων σας. Χιλιάδες αντιδράσεις. Το hashtag Europe έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από 7.000 φορές. Και να δούμε πόσα θα φτάσουμε μέχρι το τέλος της βραδιάς. Και θέλω να δω και πιο πολλούς Φιλανδούς εδώ. Χθες ε, δεν είδαμε πάρα πολλούς ε, στην διαγωνισμό της Eurovision. Για να ακουστεί λοιπόν η δική σα φωνή σήμερα, και αυτό το λέω και σε όλους τους υπόλοιπου Ευρωπαίους, μιλώντας για την δέσμευση, πολλοί από εσά μα ε, λέτε γιατί θα πάτε να ψηφίσετε στις επερχόμενες ευρωεκλογέ. ευρωεκλογές. Μας λέτε λοιπόν ε, κατά πολέμηση αλλαγή του κλίματο, για να αλλάξει η Ευρώπη και να γίνει καλύτερη, για να σταματήσει ε, ο τοξικός οθνικισμός και για να συνεχιστεί η δημοκρατία. Πώς ανταποκρίνεται λοιπόν η online κοινότητα σε αυτά τα πρώτα θέματα. Για να δούμε. Μετανάστευση. Αυτό πραγματικά έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Έχουμε ένα χρήστη από το Βέλγιο, ο οποίος λέει ότι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να υποστηρίξουν τους μετανάστες με τρόφιμα και στέγαση. Και να σας πω επίσης ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα της αλλαγής του κλίματος. Πολλοί μας στέλνετε ερωτήσεις διαφόρων ειδών για το θέμα. Από τη Γερμανία, για παράδειγμα, έχουμε μία ερώτηση προς τους υποψηφίους. Τι θα κάνετε για να καταπολεμήσετε την αλλαγή ε, του κλίματος και για την αποτροπή της κρίσης. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε πιο πολλά και από τους υποψηφίους. Για να πάμε λοιπόν και πάλι πίσω στο debate. you. Ευχαριστώ πολύ, Αναστίνα. Εξαιρετική η μετάβαση, γιατί έτσι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενό μας θέμα, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή. Βλέπετε όλοι ότι υπάρχουν χιλιάδες νέοι Ευρωπαίοι μαζί με την Κράτα Τούνμπερκ βγαίνουν στους δρόμους με τις παρασκευές για το μέλλον, Fridays for Future και το κίνημα αυτό. Κάθε εβδομάδα σχεδόν έχουμε μια νέα ε, μελέτη των επιστημόνων που ζητούν από τους πολιτικούς όπως εσείς να αναλάβουν δράση αλλά είναι πολύ ακριβή ακόμη η αποτελεσματική προστασία του κλίματος. Μπορεί να χαθούν πολλές θέσεις εργασίας από την ε, οικονομία του άνθρακα ή από την αυτοκινητοβιομηχανία, ε, ενέργεια, μπορεί να κοστίζει πιο ακριβά για τον ε, απλό πολίτη. Ερώτηση λοιπόν προς τους ε, υποψηφίου. τι θυσίες είστε διατεθειμένοι να κάνετε προκειμένου να προστατέψετε τον πλανήτη μα, κάτι περισσότερο ή τι θα μπορούσατε να κάνετε λιγότερο, παρακαλώ να δώσετε συγκεκριμένε προτάσει. Ναι, βεβαίω είναι κίνδυνο, αλλά μπορούμε να την αξιοποιήσουμε εάν το να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο αυτό ω ευκαιρία. Εκατομμύρια θέσει εργασία μπορούν να δημιουργηθούν. Για παράδειγμα, για τα τρένα υψηλή ταχύτητα. Αν φτιάξουμε ένα δίκτυο για να συνδέει τι πόλεις μα για να μπορούν να περάσουν από τα αεροπλάνα στα τρένα οι συμπολίτε μα. Αυτό είναι συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Και επίση έχουμε θέσει στόχου, έχουμε την νομοθεσία για να μεταρρυθμίσουμε τι αγορέ. Τώρα πρέπει να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα νομοθετήματα. Η τεχνολογία υπάρχει. Πρέπει να επενδύσουμε και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Και πρέπει να κάνουμε και περισσότερη έρευνα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε περισσότερη τεχνολογία. Πολλά μπορούν ήδη να γίνουν. Και εάν υπάρξει συστηματική προσέγγιση θα συμμετάσχουν όλοι μέσω των ε, προσωπικών μας επιλογών. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο οι μεμονωμένοι πολίτες μπορούν να δώσουν λύσεις. Ευχαριστώ πολύ, Μαγκρέτε Βεστάγκερ. Σκά Κέλλερ, Βεβαίως θεωρώ ότι αντιμετωπίζετε πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά, αλλά οι πράσινοι είναι διατεθειμένοι να αποτεχθούν ε, απώλεια θέσεων εργασία. Το θέμα αυτό το παίρνουμε πολύ στα σοβαρά και όλοι θα έπρεπε να το παίρνουμε στα σοβαρά γιατί είναι κατεπήγον θέμα. Έχουμε έναν και μόνο πλανήτη. Θα πρέπει να το προστατεύσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμού και να πούμε Α περιμένουμε λίγο με το κλίμα. Δεν ξέρουμε ακόμα τι να κάνουμε. Βεβαίω και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το καλό είναι όμω ότι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Τα μέσα τη πολιτική, τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε, τα ξέρουμε. Μπροστά μα είμαι. Πρέπει απλά να τα εφαρμόσουμε. Και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο δυστυχώ υποστηρίζουν οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε. Ε, ουσιαστικά καταπολεμάτε με την ψηφοφορία σα την κρίση αυτή, την αντιμετώπιση τη κρίση του αλλαγή του κλίματο και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα απώλεια βιοπικιλότητα. Είναι πραγματικά αυτό το θέμα αυτό. Τι θα κάνω εγώ, τι θα έκανα εγώ, για παράδειγμα, να σταματήσουμε τις επιδοτήσεις που βλάπτουν το περιβάλλον και που δίδονται κάθε χρόνο εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να σταματήσουμε να τα χορηγούμε Προ την κατεύθυνση αυτή και να τα χρησιμοποιήσουμε και παράδειγμα σε τεχνολογίε φιλικέ προ το κλίμα, να δημιουργήσουμε πολλέ θέσει απασχόληση. τόσες θέσει απασχόλησης που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σε τέτοιε οικονομίε, σε τέτοια οικονομία η φιλική προ το περιβάλλον και τώρα φεύγουν, πάνε στην Κίνα αυτέ οι θέσει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Φραν Τίμερμαν. πρώτο αντιπρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσατε τη βοή και τη φωνή των ανθρώπων στου δρόμου. Ναι, βεβαίω, τα άκουσα, κάθε μέρα τα ακούω όπου πηγαίνω, δέκα φορέ τη μέρα και θέλω να πω το εξή. Η Σκάκελερ είπε ξεκάθαρα λόγια. Ο κύριο Κουέ είναι από του επικεφαλεί ε, πολιτικούς στην κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον και οι τρεις μας μαζί έχουμε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι τρεις μας μαζί έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες και τους προτείνω να συνεργαστούμε για την επόμενη πενταετία για να εξασφαλίσουμε πως η προσεχή Ευρωπαϊκή, προσεχής Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέσει στο πρώτο βαθμό μελήματο το κλίμα για να δώσουμε μια απάντηση με μια συμμαχία η οποία θα πηγαίνει από τον Τζίπρα μέχρι τον Μακρόν όλη η προοδευτική οικογένεια για να θέσουμε στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών μας το κλίμα. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε φορολογία για το διοξίδιο του άνθρακα, ε, γιατί τα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν χωρίς επιβάρυνση φορολογική αυτού του τύπου που θα μπορούσε μετά να αποδοθεί ως ε, ε, πόρος στον πολίτη που έτσι θα προσαρμόσει και το σπίτι του. Μπορούμε να τα κάνουμε αυτά όλα μαζί αν συμφωνήσουμε πως μπορούμε μαζί με τα κράτη-μέλη και την υποστήριξη βέβαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει μια προσπάθεια ήδη δημιουργία συνασπισμών. Αλλά α περάσουμε τώρα σε αυτό που υποθέτω είναι η αντιπολίτευση. Γιάννη Σαχράντιλ, τι θα κάνετε για να προστατεύσετε περισσότερο το κλίμα ή θα κάνετε λιγότερα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη πριν από 30 χρόνια. Ήταν ε, η πιο μολυσμένη περιοχή όχι μόνο της Ευρώπης αλλά του κόσμου. Τώρα μειώσαμε κατά πολύ την ατμοσφαιρική ρήπανση είναι λοιπόν εφικτό, αλλά πρέπει να γίνει σταδιακά με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών. Πρέπει να είναι κοινωνικά αποδεκτό και σταδιακό το εγχείρημα αυτό. Να μην έχουμε λοιπόν υπερβολικούς στόχους. Ας δεσμευθούμε να εφαρμόσουμε αυτά που ήδη εγκρίναμε, για παράδειγμα τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, αλλά η Επιτροπή θα μπορούσε να αλλάξει για παράδειγμα τις επιδοτήσεις της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πρέπει να αντιμετωπίζουν περισσότερο τις περιβαλλοντικές ανάγκες, να επιδοτούμε περισσότερο τις μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις βιολογικής γεωργίας και όχι τις μεγάλες. Και επίσης είναι πολύ σημαντική πολιτική για το ένα εκτάριο. Θα το εξηγήσω αργότερα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ξεπεράσατε το χρόνο. Νίκο Καταρχάς ευχαριστώ τους νέους που εβδομάδες τώρα διαμαρτύρονται, εκφράζουν τη δυσφορία τους γιατί αισθάνονται ότι δεν τους ακούει κανείς. Ναι και όντως δεν τους ακούνε. Μπορεί να ακούμε πολλές ομιλίες από τους ε, Ευρωπαίους ταγούς αλλά δεν λαμβάνονται αποφάσεις. Επί παραδείγματι, δεν στρέφεται κανεί κατά των μεγάλων πολυεθνικών που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη μέχρι και 70% της παγκόσμιας ρήπανση. Δεν υφίστανται καμία κύρωση. Από την άλλη βέβαια και πρέπει να μετατοπιστεί το πρόβλημα στην, ε, στο θέμα της φορολογίας για τους πιο αδύναμους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο βλέπουμε στη Γαλλία με το Μακρόν που έχει επιβάλει τέτοια φορολογία εις βάρος των απλών πολιτών. Είναι απαράδεκτο. Έχουμε κάνει πολλά στην Ευρώπη με το πρόγραμμα Γαλιλαίος, με την Airbus γιατί, γιατί να μην προχωρήσουμε προς μια νέα πρωτοβουλία, κοινή πρωτοβουλία για το κλίμα. Μην μου πει κανεί ότι δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί 3 δισεκατομμύρια δόθηκαν για να σωθούν οι τράπεζε. Κύριε Τίμερμαν, στη δική σα ομάδα, αν δεν απατώμα, ήταν εκείνη η οποία ανακοίνωσε πω η φόρο ε, απάτη είναι ήδη πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Έχουμε πολλά χρήματα λοιπόν διαθέσιμα για να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ. Τώρα ο Μάφρετ Βέμπερ. Θα ήσασταν πιο φιλόδοξο για την προστασία του κλίματο από την ε, Επιτροπή που έχει τώρα την ευθύνη αυτή. Θέλουμε να πετύχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα είναι ουδέτερη ω προ τι εκπομπέ ανθρακά. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό προκαλεί διαφοροποίηση και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι δεσμευμένο προ το στόχο αυτό. Για το πώ ε, θα το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν ε, νομίζω ότι θα πρέπει τελικά οι χαμένοι να είναι ο κόσμος, οι συνταξιούχοι. Έχουμε πολλά μέσα με τα οποία μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Και έχουμε πολλές ανησυχίες και στην Ήπειρο και παντού. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν με έναν τρόπο που θα είναι σεβαστές οι ανάγκες όλων. Και ε, σας μιλώ ότι ήταν ο Επίτροπος ε, Κανιέτε του Ευρωπαϊκού Λογικού Κόμματος, ο οποίος παρουσίασε όλες τις προτάσεις για την ε, καταπολέμηση του αλλαγή του κλίματος. Και θα συνεχίσουμε στην πορεία αυτή. Ευχαριστώ, Μάνφρετ Βέμπερ. Κύριε Τίμερμαν, έχετε ένσταση να πω ότι έγινε μια ψηφοφορία, έγινε ψηφοφορίες μάλλον στο Κοινοβούλιο και μιλάμε για τους δεινόσαυρους του Ευρωπαϊκού Λίγου Κόμματος. Αυτά τα λένε ΜΚΟ, όχι εγώ. Και πρέπει να σας πω ότι έχω συγχαθεί πια αυτή τη δικαιολογία ότι θα βλάψει αυτό το κόσμο και το περιβάλλον. Ξέρετε, θα τους βλάψει αν δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν κάνουμε τίποτα για την αλλαγή του κλίματος, θα λάβει τεράστιες διαστάσεις. Και οι φτωχοί είναι αυτοί που θα πλεχθούν πρώτα. Δεν έχουν κάπου αλλού να πάνε. Δεν μπορούν να αποφύγουν την κρίση αυτή. Θα πρέπει να δράσουμε. Όσο πιο πολύ περιμένουμε, τόσο πιο ακριβό θα γίνει αυτό και τόσο πιο δύσκολο θα είναι και για τους φτωχούς. Ο Μάνφρετ Βέμπερ για να απαντήσει. Κοιτάξτε, πολύ σπουδαία λόγια, Φραντ Τίμερμαν και πάλι, αλλά θέλουμε συγκεκριμένε δράσει τώρα. Έχει, ώρα, έχει έρθει η ώρα για τι δράσει και σα πω ότι το σύστημα εκπομπή ε, ανταλλαγή εκπομπών ρήπων ε, αν το επεκτείνουμε στην αεροπορία, θα ήταν ένα σημαντικό βήμα αυτό. Πώ μπορούμε επίση να υποστηρίξουμε την κοινοτομία, πιστεύω, ω ε, μηχανικό, γιατί είμαι μηχανικό περιβάλλοντο. Πιστεύω στην κοινοτομία, όχι στην τιμωρία, όχι στι απαγορεύσει, όχι στα αριθμιστικά πλαίσια. Στην κοινοτομία πιστεύω. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ορίζοντα για επενδύσει ε, στην τεχνολογία για να επιλύσουμε τα προβλήματα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει χρόνος γιατί υπάρχουν πολλά άλλα θέματα. Ε, πρώτα απ' όλα έχουμε δύο ενστάσεις. Μία από τη Σκά Κέλλερ. Ναι, έχουμε σοβαρές ε, διαφορές για τα κλιματικά θέματα. Ορισμένοι απλώς μιλάνε για το κλίμα, ενώ εμείς θέλουμε κάτι να γίνει. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πολύ συγκεκριμένα ερώτηση στο Μάνφρετ Βέμπερ λέτε ότι είναι θαυμάσιο το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Γιατί η ομάδα σας τότε καταψήφισε τη μεταρρύθμισή του, ούτως ώστε να λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή δίνουμε τόσα ε, πιστοποιητικά εμπορίας ε, δωρεάν που μπορούν μετά να τα ανταλλάξουν οι μεγάλες εταιρείες χωρίς κανένα κόστος. Γιατί το καταψηφίσατε. Γιατί η ομάδα σας είναι κατά πιο αυστηρών κλιματικών στόχων. Δεν είναι πραγματική κλιματική πολιτική κάτι τέτοιο. Πριν δώσω το λόγο στον Μάνφρεντ Βέμπερ, να σας εξηγήσω ότι ETS σημαίνει σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ο κύριος Βέμπερ παρακαλώ. Ναι, γιατί το κόμμα μου προσπαθεί να υπάρξει συνολική αντιμετώπιση. Βεβαίως ορισμένοι είναι πολύ φιλόδοξοι. Οι πράσινοι για παράδειγμα ε, τονίζουν ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Αλλά εγώ συναντήθηκα με τα συνδικάτα, όχι με δικούς μου ψηφοφόρους, με σοσιαλιστές ψηφοφόρους που μου είπαν ότι αν εφαρμόσετε αυτά που προτείνουν οι πράσινοι, τότε θα χάσουμε τις δουλειές μας. Πρέπει να είναι βιώσιμα αυτά που κάνουμε. Η βιωσιμότητα, όπως λένε τα Ηνωμένα Έθνη, σημαίνουν και οικονομική βιωσιμότητα και οικονομική σταθερότητα και τεχνολογική βιωσιμότητα. Όλα αυτά πρέπει να τα συνδυάσουμε, όχι να τα αποσυνδέουμε. Ευχαριστώ πολύ. Για άλλη μια φορά όμως έχετε ένσταση από την Μάργρετ Βέσταγερ. Ναι, μια και επιμένετε ότι ο συνάρφος Μιγγέλ είναι του ΕΛΚ, θα σας θυμίσω. Δεν έκανε όμως ε, καταπληκτική δουλειά επειδή είναι του ΕΛΚ, αλλά επειδή είναι μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνάδελφος Βιολέτα Μπούρτς δεν άνοιξε το δρόμο για την ε, ε, ε, μείωση των εκπομπών του άνθρακα επειδή είναι φιλελεύθερη, αλλά γιατί συνεργαστήκαμε όλοι μαζί, γιατί έχουμε αναγνωρίσει ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα τόσο μεγαλύτερο από τη δική μας ταπεινή προσωπικότητα που πρέπει όλοι μαζί να το αντιμετωπίσουμε. Όλα λοιπόν αυτά πρέπει να τα αξιοποιήσουμε, να μην περιμένουμε άλλο. Απάντηση. Μαγκρέτε, αυτή ακριβώ ήταν και η αναρκτήρια τοποθέτησή μου. Α μην ε, διχαστούμε πάνω σε αυτό, γιατί ο στόχο μα είναι κοινό. Είμαστε στο ίδιο, ε, στην ίδια πλευρά. Και οι φιλελεύθεροι ω πολιτική ομάδα έχουν τα ίδια μελήματα για την ταχύτητα στην υλοποίηση. Το 2050 πρέπει να έχουμε βιομηχανική παραγωγή ουδέτερη ω προ τι εκπομπέ άνθρακα. Αυτό πρέπει να κάνουμε και συμφωνώ, αλλά όχι να τιμωρήσουμε του φτωχότερου με την επιβολή μια πολύ ακριβή νέα τεχνολογία. Ευχαριστώ πολύ, Μάνφρεντ Βέμπερ. Αλλά υπάρχει άλλη μία κάρτα από τον Νίκο κουε προ εσά. Θεωρώ απαράδεκτα αυτά που λέγονται εδώ. Κλείσαμε την Υψικάμινο στην Λιέγη και στη Φλωράνζ τη Χαλιβουργία πριν από 7-8 χρόνια. Τα συνδικάτα έκαναν μια σειρά από προτάσεις για ειδικού χάλιβες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την επιβίωση αυτών των εγκαταστάσεων. Φανταστείτε πόσο λιγότερη μόλυνση θα είχαμε τότε στα εδάφη μας. Θα μπορούσαμε να παραγάγουμε πολύ περισσότερα χαλιβουρικά προϊόντα. Αλλά μαζί με τον κύριο Ταγιάννη τα δώσατε στον κύριο Μιτάλ που έκλεισε τις υψικαμίνους και ο χάλιβας τώρα έρχεται από άλλες χώρες. Όχι από την Ευρώπη, μολύνοντας δυο φορές από ό,τι θα μόλυνε η δική μας χαλιβουργία. Κύριε Βέμπερ, η δική σας απάντηση. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβετε ότι βεβαίως είμαστε φιλόδοξοι ως ε, Ευρωπαίοι και ο κύριος στόχος της επόμενης Επιτροπής θα πρέπει να είναι να, πιέσει, να πείσει τον υπόλοιπο πλανήτη. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνοι μας. Χρειαζόμαστε και τους άλλους. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι φιλόδοξη σε παγκόσμιο επίπεδο, να συνεργαστεί για μια παγκόσμια λύση με τη συμμετοχή όλων για να καταπολεμήσουμε από κοινού την κλιματική αλλαγή. Αυτό θέλω να κάνω. Α, να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, ο Χουέ. Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας. Το επόμενο θέμα είναι κάτι που ανησυχεί πολλούς. Μπορεί να φαίνεται τεχνικό. Μας ανησυχεί γιατί είναι σύμβολο αδικίας. Οι πολυεθνικές όπως η Apple, η Google, η Nike πληρώνουν ελάχιστους φόρους, πολλές φορές λιγότερο από 5%. Ενώ εμείς οι πολίτες πληρώνουμε μεταξύ 20 και 40%. Οπότε, ερώτηση προς τους υποψηφίους. Ποιες χώρες κατά την γνώμη σας είναι φορολογική παράδοση, ποιες χώρες της Ένωσης και πώς θα αλλάξετε τη συμπεριφορά τους, ούτως ώστε η Amazon να πληρώνει όσα και το μικρό βιοπολείο στην πλανή πόρτα. Η Μάργαρέτε Φέσταγκερ. Τα γνωρίζω αυτά από πρώτο χέρι. Είσαστε πολύ γενναιόδωρο όταν λέτε ότι κάποιε πληρώνουν μόνο 5% διότι γιατί κάποιε εταιρείε πληρώνουν 0,05% φόρου, όπω είδαμε στην περίπτωση τη Apple. Όντω, λοιπόν, πολλά έχουμε να κάνουμε μπροστά μα. Αυτό που είδαμε είναι ότι τα κράτη-μέλη αλλάζουν ε, στις φορολογικά στο καθεστώτα στην Ιρλανδία, στην ε, Μάλτα, στην Κύπρο, ε, παντού, γιατί υπάρχει ένα κύμα αλλαγών. Έχουμε αλλάξει την νομοθεσία παντού, αλλά χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Ψηφιακή αφρολόγηση γιατί πολλές από αυτές τις εταιρείε διαφεύγουν και οι πιο πολλές επιχειρήσεις πληρώνουν τους φόρους τους. Αυτό είναι άδικο. Και δεύτερον, Χρειαζόμαστε να υπάρχει ένα κατώτατο επίπεδο σε ό,τι αφορά την ε, φορολόγηση των επιχειρήσεων. Γιατί λιντάλλω όλοι θα προσπαθούν να πάνε πιο κάτω. Και θα πρέπει επίση να δούμε και στι ε, εταιρείε, στι κοινωνίε να υπάρχει σωστή και δικαιοσύνη. Ναι, λοιπόν, οι χώρε που αναφέρατε είναι φορολογική παράδειση. Για μένα, φορολογικό ε, παράδεισο είναι ένα τόπο όπου όλοι πληρώνουν του φόρου του ευχαριστώ, ευχαριστώ Μάρκετ Βεστάιερ. Σκά Έλερ είστε το ίδιο αισιόδοξοι με την κυρία Βεστάιερ. Ναι, ελπίζω πράγματι, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πραγματικό σκάνδαλο Είπατε ότι είναι πολύ χαμηλή η φόρη που πληρώνουν οι μεγάλες αυτές επιχειρήσεις, οι πιο ισχυροί δηλαδή της κοινωνίας, διαφεύγουν των ευθυνών τους και αυτό κοστίζει τόσα πολλά στον κοινό φορολογούμενο από χρήματα που δεν έχει για τα σχολεία, για τα νοσοκομεία, για την καλή εκπαίδευση και ε, δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν έχει κέριο, κέρια σημασία η φορολογική δικαιοσύνη. Για την κοινωνική δικαιοσύνη χρειάζεται λοιπόν φόρος για τις ψηφιακές, για τις μεγάλες μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν εύκολα να διαφύγουν τις ε, φορολόγησης και ένα ελάχιστο ποσοστό για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται και διαφάνεια και αυτό πρέπει να ισχύει για όλες τις εταιρείε. Ήδη υπάρχουν κοινοί ε, κανόνες που έχουν εγκαθιδρυθεί, που έχουν επιβληθεί. Πρέπει να γνωρίζουμε τι ε, κομμάτια παραγωγής ε, επιχειρήσεις ε, θηγατρικές κτλ. έχει μια πολυεθνική σε διάφορες χώρες ενώ έχουν κάποιοι ψηφίσει για εξαιρέσει στη διαφάνεια. Η διαφάνεια δεν μπορεί να ισχύει για κανέναν. Ευχαριστώ πολύ Σκάκελα. Και τώρα, Φραντ Τίμερμαντ. Αναφέρθηκε ήδη η χώρα σα. Είναι φορολογικό παράδεισος, Τίμερμαντ. Ναι, είδαν τι πρόκειται να συμβεί και επιτέλους ε, ε, ε, αποφάσισαν να αλλάξουν. Συμφωνώ με τη Μαγκρέτε Φεστάκερ. Χρειαζόμαστε ένα ελάχιστο επίπεδο εταιρικού φόρου παντού στην Ευρώπη. Α πούμε 18% ελάχιστο ποσοστό, ελάχιστο φορολογικό συντελεστή. Οπότε οι χώρε μπορούν να επιβάλλουν μεγαλύτερο εταιρικό φόρο, αλλά όχι λιγότερο. Επίση, έχει αλλάξει τόσο θεμελιωδώ η οικονομία. Είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Οι εταιρείε έχουν βρει τρόπου να πληρώνουν καθόλου φόρου. Έχει δίκιο η Μαγκρέτε. Οι μεγάλες επιχειρήσεις σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρώνουν φόρο. Θα πρέπει λοιπόν να ρωτάμε την Αλέξα, η Amazon πότε θα πληρώσει φόρους. Ε, και επειδή έχετε ακόμη 20 δευτερόλεπτα, 18% προτείνεται. Πώς η Ιρλανδία θα συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο. Τίμερμαντς, ναι, μα βλέπουν ότι στην ουσία μακροπρόθεσμα θα θίξει την οικονομία τους έχουν τι ε, τεράστιε αποθήκε όπου δεν δουλεύει κανένα. Αυτό δεν ε, βοηθάει καμία οικονομία. Μπορούμε να του πείσουμε όλου να ακολουθήσουν αυτή την οδό του ελάχιστου εταιρικού φόρου. Είναι δείγμα φορολογική αλληλεγγύη. Μπορούμε να πείσουμε και τη δική μου χώρα, πιστεύω. Ευχαριστούμε, Φραν Τίμερμαν. Ε, Γιάνν Ζαχάντιλ, τι έχετε να πείτε για την φορολογική πολιτική. Καταρχάς να πω ότι θα υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ μας κατά πάσα πιθανότητα γιατί θεωρώ ότι τα κράτη έχουν δικαίωμα να φορολογούν τι επιχειρήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτο. Μπορεί κάποιοι να ήθελαν να είναι κράτο. Στην περίπτωση αυτή, καταλαβαίνω ότι ζητούν ευρωπαϊκού φόρου. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω παρόλα αυτά ότι φυσικά η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή θα πρέπει να απαγορεύεται και έχουν ε, γίνει σωστά βήματα. Υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ε, κύκλο εργασιών πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ είτε πληρώνουν φόρους εδώ ή εκεί. Άρα μπορούμε να εντοπίσουμε εύκολα αυτούς που δεν πληρώνουν φόρους και θα πρέπει να υπάρξει φορολόγηση σε εθνικό επίπεδο. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει φορολόγηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και παρεπιπτόντω, να πω ότι η Επίτροπο Φεστάκερ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ για να δημιουργήσει ίσου όρου ανταγωνισμού και για να προσπαθήσει να πετύχει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ Γιάννη Ζάγραντελ. Νίκο Κουέ, συμφωνείς ότι η Ευρώπη δεν έχει ε, δουλειά να καθορίζει φορολογικούς συντελεστέ. Καθόλου μάλιστα. Στην Ευρώπη υπάρχουν ε, ορισμένες περιοχές όπου δεν υπάρχουν ε, σχολεία, δεν υπάρχουν νοσοκομεία, δεν υπάρχουν συγκοινωνίες. Δεν υπάρχουν ε, δημόσιες παροχές. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία δυνατότητα οι φόροι να βοηθήσουν ε, τον πληθυσμό αυτών των περιοχών. Πόσο καιρό τώρα συζητάμε για κάποια εναρμόνιση για να αποφύγουμε το φορολογικό dumping που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτοί πολλά χρόνια τώρα ενώ είναι στην κυβέρνηση αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν κάνει κάτι το ουσιαστικό. Πρέπει να κάνουμε κάτι το πραγματικά ουσιαστικό για την φοροαπάτη. 850 δις λέγεται ότι είναι η φοροδιαφυγή. Πόσα σχολεία, πόσα νοσοκομεία θα μπορούσαμε να φτιάξουμε. Και επίσης να υπάρξει η ελάχιστη σοβαρότητα. Αυτοί που καταγγέλουν τα σκάνδαλα και την φοροδιαφυγή να προστατεύονται και όχι να καταδικάζονται Ευχαριστώ πολύ, Νίκο Κουέ. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ. Ήμουν ε, περήφανο στου Ευρωπαίου όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί κατά τη Ιρλανδία. μαγκρέτα εσεί και ο Ζων Κλοντ Γιούγκερ για να εξασφαλίσουν ότι θα πλήρωναν όσο του αναλογούσαν για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε. Να χρησιμοποιούμε την οικονομική μα ισχύ και το ρυθμιστικό πλαίσιο για να πληρώνουμε όλα αυτά που πρέπει. Και θα πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε του φορολογικού παραδείσου. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα από την φορολόγηση αυτή για να διαμορφώσουμε, να μεταρρυθμίσουμε την διαδικασία τη ψηφιοποίηση. Έχουμε κοινέ ιδέε. Το θέμα όμω είναι πώ θα τα πετύχουμε αυτά. Και γι' αυτό θα πρέπει να σημειωθούν αλλαγέ σε κάποιου ε, τομεί τη φορολογία ε, από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία στη λήψη αποφάσεων. Και πραγματικά πιστεύουμε σε αυτή την προσέγγιση γενικώ πώ Πιστεύω στον φορολογικό ανταγωνισμό, αλλά σε ειδικού τομεί, όπω είναι για παράδειγμα η ψηφιακή φορολόγηση, χρειαζόμαστε έναν κοινό ευρωπαϊκό δρόμο. Ευχαριστώ, Μάνφρετ ε, Βέμπερ. Θέλω να επισημάνω ότι στο στάδιο αυτό τη συζήτηση έχετε όλοι χρησιμοποιήσει τι πρώτε κάρτε ένσταση, αλλά σα μένει η δεύτερη για τον καθένα κάρτα ένσταση προ του συνυποψηφίου. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Ε, καυτά θέματα αυτά του περιβάλλοντος, της φορολογίας. Αναστήνα, τι λέει ο κόσμος. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στον κόμβο της, ε, των μέσων ψηφιακή ενημέρωση. Πραγματικά ακούγεται η φωνή σα ε, στο hashtag Tell Europe. Σα ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Για να σα δώσω μια καλύτερη εντύπωση για το τι λέει ο κόσμο online. Να σα δώσω, να σα δείξω ε, τι βασικέ έννοιε που χρησιμοποιούνται. Το κλίμα, η πράσινη, ανάπτυξη. Οι πιο βασικές ε, έννοιες που χρησιμοποιούνται. Climate και green. Όπως ε, βλέπετε, πολλοί θέλουν να γνωρίσουν και πιο ε, καλά τους υποψηφίους και να γνωρίσουν και πιο πολλά πράγματα για τις εκλογές, να ενημερωθούν και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εκλογές θα λάβουν χώρα 26 με 28 Μαΐου. Ένα άλλο βασικό λοιπόν θέμα είναι το θέμα της ισότητας των φύλων, gender equality. Ένας χρήστης θέλει να μας πείτε πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα της διαφοράς μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Με την ε, άνοδο των προσκεπτικιστών και των λαϊκιστικών κινημάτων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, κάποιοι χρήστες εξέφρασαν μια γενική δυσαρέσκεια και έλλειψη εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα tweet από τη Γερμανία να δούμε, το οποίο θεωρώ συνοψίζει πολύ εύστοχα το αίσθημα πολλών από εσάς. Θεωρούν λοιπόν πολλοί ότι δεν ε, ξέρουν αρκετά καλά, δεν εξηγείται αρκετά καλά τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στείλτε μας λοιπόν ε, τα σχόλιά σας στο hashtag Tell Europe και να συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, Αναστίνα. Και τώρα να περάσουμε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έναν κόσμο όπου κυριαρχούν οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα. Όλο και πιο συχνά η Ένωση βρίσκεται σε αντιπαράθεση με αυτέ τι μεγάλε δυνάμει, είτε για τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, είτε για το Nord Stream 2, είτε για το ελεύθερο εμπόριο. Επανειλημμένα, ο πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ απειλεί για νέου δασμού επί ευρωπαϊκών προϊόντων. Είναι πολύ ευρύ το θέμα. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η δική σας ε, θέση. Οπότε, ερώτηση. Για να συμφωνήσουμε με τον Ντόναλτ Τραμπ που θα είναι μάλλον καθήκον ε, της επόμενης Επιτροπής για να αποφύγουμε τη ζημιά στην ευρωπαϊκή οικονομία. Είστε διατεθειμένοι να ανοίξετε τις ευρωπαϊκές αγορές στα αμερικανικά γεωργικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων και των γενετικά τροποποιημένων όπως από ό,τι φαίνεται απαιτεί ο Τραμπ. Πρώτη απάντηση από τη Σκά Κέλλερ, παρακαλώ. Όχι, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και λίγο παραπέρα. Να σκεφτούμε ποιο ρόλο θέλουμε να τερματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο. Και νομίζω ότι θα είχαμε σημαντικό ρόλο να παίξουμε. Ποιο θα είναι ο ρόλο αυτό, και θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι εδώ. Και πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι δύναμη ειρήνη και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Εδώ μπορούμε να αποστείλουμε ένα πραγματικά ηχηρό μήνυμα και πραγματικά να κάνουμε κάτι. Γιατί κάνουμε πολλά πράγματα. Είμαστε ο μεγαλύτερο δωρητή για τα δικαιώματα, τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Αλλά δεν είμαστε συνεκτικοί, δεν, είμαστε, δεν μιλάμε με μία φωνή. Θα πρέπει να πούμε ότι ω Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνουμε και όπλα στου δικτάτορε που καταπιέζουν του λαού. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεκτικοί στην αντίδρασή μα. Να σταματήσουμε να αποτελούμε και ε, για παράδειγμα, να αφήνουμε τους δικτάτορες να βάζουν τα χρήματά τους στις ευρωπαϊκές τράπεζες και αυτό να το κάνουμε παντού και πάντα. Ευχαριστώ, Όσκα Κέλλερ. Φρανς Τίμερμανς. Τι στάση θα τηρήσετε απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα. Απάντηση. Μα είμαστε πολύ ισχυροί ω Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν έχουμε ηγέτε στην Ευρώπη που είναι οι καλύτεροι φίλοι του Βλάντιμιρ Πούτιν και πάνε και του στάνε λεπτά και μετά πάνε στον Τραμπ να του στήσουν ακρόαση, όταν ξέρουν ότι αυτό προσπαθεί να διαλύσει την Ευρώπη, ενότητα πώ θα εξασφαλίσουμε. Πρέπει να αντιληφθούμε τι διακυβεύεται εδώ για μα, του Ευρωπαίου. Είναι η πρώτη φορά στην Ευρώπη, στην ιστορία, που υπάρχει Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίο θεωρεί πω είναι προ το συμφέρον του να διαλύσει την Ευρώπη. Πρέπει να αντισταθούμε λοιπόν, να αντισταθούμε με τι αξίε μα στον κόσμο κόσμο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ενότητα, χρειάζεται να πιστούν οι πολιτικέ εκείνε δυνάμει οι οποίε θεωρούν ότι ο Πούτιν είναι ο καλύτερό του φίλου, από το Φαράζ μέχρι το Σαλβίνη, τον Στράχα. Όλοι αυτοί πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν έχουν ω κύριο μέλημα το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων, να υψώσουμε τον παράστημα στον Τραμπ, στον Πούτιν και αν δεν αντιληφθούμε τι διακυβεύεται εδώ, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ. Μάνφρετ Βέμπερ. Μπορούμε να λέμε απλώς όχι κάθε φορά που μας πιέζει ο Τραμπ. Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί είναι, ο Αμερικανικός λαός είναι πάντα φίλοι μας. Έχουμε πολλές κοινέ αξίες, ε, ελευθερία του τύπου, ανεξάρτητη δικαστική εξουσία, ισότητα των φίλων και δημοκρατία γενικά. Έχουμε πολλά κοινά. Γι' αυτό δεν στρεφόμεθα κατά του Αμερικανικού λαού, αλλά αυτά που κάνει ο Λευκό Οίκο φυσικά δεν μα βρίσκουν σύμφωνου. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σαφεί και ανοιχτοί. Στον Αμερικανικό πρόεδρο θα του πω για παράδειγμα για τα βιομηχανικά προϊόντα, για το εμπόριο, α καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά μόνο αν θέλετε ισότητα. Αν θέλει να μα πιέσει, θα αντισταθούμε. Γι' αυτό η ενότητα είναι η ισχύ μας. Χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό για να μπορούμε να συζητήσουμε. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι δύσκολο να αντιδράσουμε διότι χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο. Πρέπει να περάσουμε σε πλειοψηφία γιατί αλλιώ δεν μπορούμε να αντιδράσουμε όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Μόνο εάν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή Ευρώπη στην παγκόσμια σκηνή. Ευχαριστώ, Μάνφρετ Βέμπερ. Νίκο Κουέ. Τι λέτε εσείς, τι μπορούμε να έχουμε σαν δυνατότητες απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα. Απάντηση. Πιστεύω ότι οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών αποδυναμώνουν την Ευρώπη. Γιατί δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στου εταίρου μα κοινωνικέ και περιβαλλοντικέ ρήτρε και προδιαγραφέ. Είναι κρίμα. Αν κοιτάξουμε στο σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών, αποτελούμε τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, την πιο ισχυρή. Δεν μπορούμε όμω δυστυχώ να εξασφαλίσουμε το σεβασμό του επίπεδου ζωή μα και διαβίωση. Οι ελεύθερε συναλλαγέ σημαίνουν ταυτόχρονα πω αποδίδεται η ε, εξουσία σε μια δικαιοσύνη ιδιωτική χαρακτήρα και η οποία θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα κράτη σε σχέση, εκθέτει τα κράτη δηλαδή έναντι αυτής της δικαιοσύνης. Παράδειγμα, η Αίγυπτος με το Βεόλια ε, τέθη σε αμφισβήτηση ο ελάχιστος μισθός με την εταιρεία Βεόλια λόγω αυτών των ιδιωτικών διαιτητικών δικαστηρίων. Απαραίτητο λοιπόν είναι να συζητήσουμε οι Ευρωπαίοι για όλες αυτές τις συμφωνίες γιατί πλήττουν και τον Γεωργό και τη βιομηχανία ολόκληρο τον κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ Νίκο Κουέ. Κύριε Ζαχράντιλ, θα συζητούσατε για συμφωνία για γεωργικά προϊόντα. Καταρχάς, πρέπει να πω, το εμπόριο για μας, για την Ευρώπη, αποτελεί τη, βασική μηχανή α, οικονομικής ανάπτυξης και θεωρώ ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με, την Ευρωπα... με την ε, Συνωμένες Πολιτείες, γιατί το διατελετικό εμπόριο αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία ανεξάρτητα από το ποιο είναι ο εκάστοτε Αμερικανό πρόεδρο. Αλλά δεν είναι και μοναδική αγορά, υπάρχουν και άλλε αγορέ και ήμουν ως αντιπρόεδρος της ε, Επιτροπής Εμπορίου που ε, είχαμε την ε, συμφωνία εμπορίου με την Κίνα, η μεγαλύτερη ζώνη ελευθερών εμπορίου στον κόσμο με τεράστιο συνολικό Είναι καλό αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουμε και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε καιρούς αύξησης πρωτοταυτισμού για να υπερασπιστούμε το ελεύθερο εμπόριο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και τις χώρες της Ασίας, γιατί εκεί είναι το μέλλον, το οικονομικό μέλλον του κόσμου. Ευχαριστώ, Γιάννη Ζαχράντιλ. Μάγκρετ Φέσταια. ως Επίτροπος Ανταγωνισμού εσείς, είχατε να αντιμετωπίσετε αυτές τις άλλες μεγάλες χώρες του κόσμου, τι έχετε να πείτε. Ναι, η Ευρώπη θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ισχυροί και απαιτητικοί. Είμαστε η μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερος χώρος εμπορίου και έχουμε συμφωνίες με 80 χώρες. Θα μπορούσαμε να είμαστε και μάλιστα πιο σκληροί. Εάν δίνουμε πρόσβαση στις αγορές, τις δικές μας, θα πρέπει να έχουμε και εμείς πρόσβαση σε άλλες αγορές και πρέπει να βοηθάμε και τις επιχειρήσεις μας όταν αντιμετωπίζουν αθέμητο ανταγωνισμό εκτός Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε πιέσει μέχρι στιγμή από αυτόν. Και... Κοιτάξτε, θέλετε να σταματήσω ε, ε, αυτό, αυτό, ε, αυτός ο τρόπος που φαίνεται από τον τρόπο που με κοιτάτε. Α, α, κοιτάξτε. Δεν υπάρχει πια η παλιά αντίληψη για το ελεύθερο εμπόριο. Λέμε ότι το εμπόριο πρέπει να βασίζεται στι αξίε που ανταλλάσσονται. Γιατί έχουμε ε, διάφορα θέματα για το ρόλο των ανθρώπων, για την ε, μεταχείριση των ζώων. Γι' αυτό οι συμφωνίε μα με την Ιαπωνία και τον Καναδά είναι καλέ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε το εμπόριο να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεων εργασία. Ευχαριστώ, Μαρκαρέτε Βεστάγκερ. Άλλη ένσταση από τον Νίκο Κουέ. Αλλά δεν ξέρουμε ποιον θέλετε, σε ποιον θέλετε να απευθύνετε αυτή την ε, κάρτα. Στον κύριο Τίμερμανς, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ξέρω ότι η πολιτική του οικογένεια, τουλάχιστον στην Βαλονία του Βελγίου, εκδήλωσε πολλές αντιδράσεις κατά αυτής της συμφωνίας της ΣΕΤΑ με τον Πολ Μανιέτ, πρόεδρο της ε, τοπικής κυβέρνησης της Βαλονίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να αντιληφθούμε πώς είναι δυνατόν εάν υπάρχει μια σειρά από οράματα για το μέλλον μέσα από αυτές τις συμφωνίες, αυτές οι συμφωνίες τελικά να τυχάνουν διαπραγμάτευσης έξω από τον έλεγχο των κρατών σε ένα έξω ευρωπαϊκό χώρο ε, κλειστό και έξω από τη δικαιοσύνη. Δεν έχουμε αρκετά ισχυρού θεσμούς ευρωπαϊκούς και δημοκρατικούς ώστε τα θέματα αυτά να συζητηθούν παρουσία του Ευρωπαίου πολίτη και να γίνει ο διάλογος. Απάντηση. Σα πω αμέσω. Αυτό που έκανε ο Πολ Μανιέτ, αυτό που κάνατε μαζί του, είχε τεράστια επίδραση στη φύση τη ε, συνθήκη. Και το αναφέρατε, αναφέρατε το θέμα τη ιδιωτική διαιτησία. Τώρα είναι πολύ πιο έντονο ο δημόσιο χαρακτήρα αυτή τη διαιτησία και το επικύρωσε μάλιστα αυτό και με απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Δική σα δράση λοιπόν με τον Πολ Μανιέτ μα ε, βοήθησε να πιέσουμε προ μία περισσότερο δημόσιου χαρακτήρα διαιτησία ανοιχτή δηλαδή. Ωστόσο δεν έχουν όλα αριθμιστεί. Δεν θέλουμε να γίνονται οι ρυθμίσεις αυτές μέσα σε διαπραγματεύσεις απόρριτες για κάτι το οποίο είναι κάτι που πρέπει να γίνεται δημόσια. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς, ε, Μάνφρεντ Βέμπερ, έχετε σηκώσει την κάρτα σας προς ποιον. Στην κυρία Σαχραντήλη, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα αυτό που είπατε. Έχουμε 36 εκατομμύρια ε, θέσει απασχόληση σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει να κάνει με το εμπόριο. Είμαστε μια ήπειρο του εμπορίου. Η οικονομία μας λοιπόν βασίζεται στο εμπόριο και γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι αριστεροί και οι σοσιαλιστές δεν είναι σταθεροί. Γιατί δεν λένε ναι, να χρησιμοποιήσουμε το εμπόριο για να είναι καλύτερος χώρος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται για παράδειγμα με την παιδική εργασία σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν χρησιμοποιούμε την μόχλευσή μας για να την καταργήσουμε. Γιατί λοιπόν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το θέμα στην αριστερά. Νίκο Κιουέ, θέλετε να απαντήσετε. Ναι, Λόγια πάλι. Λόγια πάλι, αλλά στην πράξη υποβιβάζεται τις κοινωνικές προδιαγραφές ε, τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές για να επιτρέψετε να εγκαθιδρυθούν αυτές οι συμφωνίες χωρίς μηχανισμούς, χωρίς ακόμη και υπηρεσίες ευρωπαϊκές οι οποίες θα μπορούσαν να επαληθεύσουν την διαφύλαξη του επίπεδου ζωής των Ευρωπαίων. Πάντα κάνετε ομιλίες οι οποίες τελικά δεν ε, οδηγούν στην πράξη, στην διαφύλαξη του ευρωπαϊκού επίπεδου διαβίωσης. Σας υπενθυμίζω κύριε Βέμπερ ότι έχουμε πολύ σημαντικέ αρχές, έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους που εργάζονται στην εσωτερική οικονομία οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις συμφωνίες διεθνούς εμπορίου, τις δικές σας συμφωνίες, ε, εξολοθρεύεται αυτή την εσωτερική οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, Σκακέλερ. Και εμένα μου ζητήσατε να απαντήσω και έχω και εγώ φαντάζομαι 30 δεύτερα. Πιστεύω ότι το εμπόριο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά πρέπει να το δούμε ω εργαλείο για την επίτευξη ενό στόχου, ένα μέσο για την επίτευξη του στόχου και όχι ω αυτό σκοπό. Γιατί αυτό φαίνεται ότι γίνεται. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν τι γίνεται στο εμπόριο. Για παράδειγμα, φιλελευθερωποίηση, απελευθέρωση των ε, υπηρεσιών για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αν ε, χρησιμοποιούμε πρωτεσίλε από άλλε χώρε, Πραγματικά αυτό δεν είναι σωστό για τη δημιουργία ενός πραγματικά πολυμερού συστήματος ε, ανάπτυξης. Άρα ποιος είναι ο σκοπός σε κάθε περίπτωση να κοιτάμε. Σας ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ κύριε Ζαχράντιλ, εσείς σε ποιον θέλετε να σηκώσετε την κάρτα σας. Ναι, ερώτηση προ τον κύριο Βέμπερ, γιατί με εξέπληξε λέγοντα ότι είναι υπέρ τη ε, ειδική πλειοψηφία σε θέματα εξωτερική πολιτική. Εγώ πιστεύω ότι η εξωτερική πολιτική είναι θέμα όπου τον κύριο ρόλο παίζουν τα εθνικά συμφέροντα. Από την έννοια τη εθνική κυριαρχία. Για παράδειγμα, για τη Λιβύη. Η Ιταλία στηρίζει τον στρατηγό Χαφτάρα, ενώ η Γαλλία Α, όχι, αντίστροφα. αντίστροφα. Η μία από τι δύο χώρε, εν πάση περιπτώσει, υποστηρίζει αυτόν τον ε, φύλαρχο, ενώ η άλλη χώρα στηρίζει την ε, νόμιμη κυβέρνηση στην Τρίπολη. Πώ είναι δυνατόν να υποχρεώσετε μέσω πλειοψηφία η χώρα ή κάποια χώρα να αλλάξει στάση. Δεν λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Θα υπάρξει ακόμη περισσότερο διχασμό μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Βέμπερ. Μα το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, είναι αναγκαίο. Μα βλέπετε ακριβώ τι συμβαίνει στη Λιβύη. Βλέπετε τι γίνεται στην Βενεζουέλα. Χρειαστήκαμε τέσσερι εβδομάδε για να καταλήξουμε σε μια κοινή ευρωπαϊκή θέση κατά του κομμουνιστικού καθεστώτο Μαδούρο. Τέσσερι εβδομάδε. Γιατί κάποιοι από την Ελλάδα και την Ιταλία αντιτίθεντο. Αυτή δεν είναι η Ευρώπη την οποία επιθυμώ. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίζει τι αξίε μα. Ελευθερία, δημοκρατία, κράτο δικαίου. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν λαμβάνουμε αποφάσεις μέσω πλειοψηφία. Έτσι θα έχουμε ισχυρή Ευρώπη για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Άλλη ένσταση από την Μαγκρέτε Βέσταγκερ. Για προς ποιον Θέλω απλώς με τη ΣΚΑ Κέλλερ να συζητήσουμε τα θέματα του εμπορίου. Γιατί υπάρχει νομίζω και μια διάσταση κλιματικής αλλαγής εδώ. Έχουμε μια σλοβενική επιχείρηση, παραδείγματι, πολύ γνωστή γιατί έχει αναπτύξει οικολογικά αεροπλάνα. Έχουμε πολλές επιχειρήσεις ευρωπαϊκές ε, οι οποίες ε, αναπτύσσουν τις ανεμογεννήτριες ή ασχολούνται με την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων. Πώς θα τα εξαγάγουμε όλα αυτά τα προϊόντα μας, αν δεν υπάρχουν τέτοιε συμφωνίε που είναι μέσα για τι εξαγωγέ και βέβαια πρέπει να αναζητούνται πάντα οι καλύτερε δυνατέ λύσει. Αυτό το γνωρίζουμε ήδη απάντηση. Ναι, συμφωνώ και δεν θέλουμε να διακοπεί ή να πάψει το εμπόριο, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε ακριβώ το παράδειγμα, το υπόδειγμα τη κλιματική διάσταση που αυτή τη στιγμή πουθενά δεν αναγράφεται σε αυτέ τι συμφωνίε. Πουθενά δεν λέγεται ότι πρέπει να υπολογίζονται οι εκπομπέ και οι ρήποι, ε, το διοξίδιο του άνθρακα, η Συμφωνία των Παρισίων. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να ακούγονται σαν ε, διακοσμητικά λόγια, αλλά έχουν ουσία. Πρέπει η διάσταση τη Συμφωνία των Παρισίων να μπαίνει σε κάθε συμφωνία εξωτερική εμπορικών συναλλαγών και αυτό το έχουμε διεκδικήσει. Δεν έχουμε εξασφαλίσει ακόμα την ε, υποστήριξη από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά συνεχίζουμε γιατί πρέπει να μπει το περιβάλλον και στις εμπορικές ε, συμφωνίες. Uh, Ευχαριστώ. Όλοι έχετε τώρα ε, πλην του Φραν Τίμερμαντς εξαντλήσει τις κάρτες ένστασης. Εσείς έχετε ακόμα μία. Την περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και τις απαντήσεις σας. Και το τελευταίο θέμα, ε, η ομάδα θεμάτων, είναι η όλο και πιο έντονη αίσθηση που έχουν πολλοί ε, πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί πια ε, όπως πριν. Οι Βρετανοί ψήφισαν να αποχωρήσουν από την Ένωση. Στην Ουγγαρία ο Βίκτορ Όρμπαν κερδίζει εκλογές με σύνθημα «Σταματήστε τις Βρυξέλλες». Αντίστοιχα και στην Ιταλία ο Ματέο Σαλβίνη. Οι ευρωπαϊκές αξίες είναι υπό απειλή ήδη υπάρχει μια διαδικασία για παραβίαση τη νομοθεσία κατά της Πολωνίας και Ουγγαρίας, του κράτους δικαίου καλύτερα ε, και θα ακολουθήσουν και άλλες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και η προσέλευση στι ευρωεκλογέ μειώνεται διαρκώς. Ερώτηση λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα του ευρωσκεπτικισμού. Ποια είναι η ευθύνη δική σα, Σκάκελα. Νομίζω ότι το θέμα είναι πιο μεγάλο, πιο ευρύ. Το θέμα είναι ο εθνικισμό, ο οποίο διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δυνάμει που θέλουν να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και που επίση δεν αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Και προφανώ πολλά θα πρέπει να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε. Καταρχά, να μην του δώσουμε πάρα πολύ χώρο, θεωρώ. Δεν είναι νόμος της φύσης ότι θα πρέπει να διωγγώνονται ως δυνάμεις στις ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι μας ως Ευρωπαίοι συμμετέχουμε στην απόφαση αυτή, στο πόσο χώρο δίνουμε στι ευρωεκλογέ, για παράδειγμα, στι εθνικιστικέ αυτέ φωνέ και στα πολιτικά κόμματα. Θα πρέπει να πάρουμε αποφάσει. Συνεργαζόμαστε με τι εξτρεμιστικέ αυτέ δυνάμει. Δυστυχώ υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Αυστρία. Το ΕΛΚΑ ε, υπάρχει συνεργασία με τα κόμματα αυτά. Έχουμε το θέμα του Ορμπάν ε, που δεν έχει επιληθεί. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το κατά πόσον αποστιωποιούμαστε επαρκώς από τέτοια κόμματα. Ευχαριστώ Σκάκελε. Φρανς Τίμερμανς. Ποιο ποσοστό ευθύνη έχετε κι εσείς είτε αφορά την πολιτική είτε τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνεται για τη δράση τη Επιτροπή. Θέλω να είμαι σαφή, λέει ο κύριο Τίμερμαντ. Ορισμένοι που ψήφισαν για το δικό μου κόμμα και ορισμένα κόμματα που εκπροσωπούνται εδώ ψηφίζουν για εθνικιστικά ορισμένε φορέ και πολύ ακραία κόμματα. Και αυτό είναι δική μα ευθύνη. Δεν του πείσαμε του ψηφοφόρου να συνεχίσουν να μα ψηφίζουν. Φαίνεται ότι πιστεύουν αυτά που λένε τα άλλα αυτά κόμματα. Αλλά θα του απογοητεύσουν τελικά αυτά τα κόμματα. Κοιτάξτε τι διχασμό έχει προκαλέσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το Brexit. Είναι σαν το Game of Thrones ε, υπερβολικό. Λόγω αυτής της πολιτικής του διχασμού έχουμε λοιπόν συλλογική ευθύνη. Πρέπει να κάνουμε προτάσεις προς τους συμπολίτε μας που να τους πείσουν ότι πρέπει να επανέλθουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και να στηρίζουν τα κόμματα που προσωπούνται εδώ που έχουν επικοδομητικές προτάσεις για το μέλλον. Αυτή είναι η μόνη διέξοδος. Ναι, είναι ευθύνη μα, αλλά έχουμε και λύσεις που τις συζητήσαμε σήμερα. Ο καθένας έχει τις ιδέες του. Πρέπει να συζητήσουμε μαζί για να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκή ενότητα για να λύσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ, Φρανς Τιμερμάν. Στην Τι έχετε να πείτε. Υπήρχε ενότητα ευρωπαϊκή αυτή τη στιγμή αποδιαρθρώνεται η Ευρωπαϊκή Ενότητα και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να αποδιαρθρωθεί η Ευρωπαϊκή Ενότητα γιατί επευλήθη με άνευ προηγουμένου βιαιότητα, λιτότητα κατά των χωρών του Νότου, κατά των Ευρωπαίων πολιτών και δεν είναι αξιοπερίεργο το ότι κάποια στιγμή κάποιε ψήφοι στρέφονται προς τα άκρα. Και βεβαίω δεν μπορώ να συγχωρήσω αυτά τα οποία προσπαθούν να κάνουν οι φασίστε στην Ιταλία, την Ουγγαρία και αλλού. Αλλά πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Ή θα κάνουμε την επιλογή των αγορών και συστηματικά θα ακολουθούμε του νόμου, τον νόμο τη αγορά ή θα κάνουμε την επιλογή του πολίτη, για τον πολίτη, για αυτούς που μένουν στην Ευρώπη. Σε αυτούς πρέπει να στραφούμε, σε αυτούς πρέπει να δώσουμε λύσεις. Και εδώ, ενώ έχουμε μειώσει τις ε, συντάξεις τους, έχουμε αυξήσει το όριο σταξιοδότησης, έχουμε μειώσει τις δημόσιες δαπάνες, είναι προφανές ότι αυτή η δυσφορία θα οδηγήσουν ανθρώπους που βρίσκονται σε πρόβλημα στη σκέψη ότι θα τους δώσουν τη λύση αυτή η ακραία. Και αυτά τα έχετε προξενήσει εσείς με αυτές τις πολιτικές Ευχαριστώ. Ε, έληξε ο χρόνος σας. Λοιπόν, η Σκά Κέλλερ και ο Φρανς Τίμερανς έχουν τις δύο τελευταίες κάρτες ένστασης. Αλλά τώρα να δώσω το λόγο στο Μάνφρετ Βέμπερ. Το κόμμα μου, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Χριστιανοδημοκράτε εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι από τα ιδρυτικά κόμματα τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ότι έχει επανέλθει ο εθνικισμό και ο εγωισμό στην Ήπειρο μα. Αλλά στις 26 Μαΐου θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτούς που θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη μας, θα πρέπει να προσπιστούμε την Ευρώπη μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δύο στοιχεία έχουμε. Θέλουμε να κάνουμε την Ευρώπη δημοκρατική. Σε ό,τι αφορά το Brexit, το βασικό μήνυμα των υπερμαχών του Brexit ήταν ότι θέλουμε την επικυριαρχία μα πίσω. Ο κόσμο δεν αισθάνεται ότι είναι δική του η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αισθάνονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μέρο ε, όπου λαμβάνονται αποφάσει για το μέλλον τη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια πιο δημοκρατική λοιπόν Ευρώπη. Κατά δεύτερον, ένα μηχανισμό χρειαζόμαστε για να προασπιστούμε τι αξίε μα, οι οποίε αμφισβητούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε έναν ανεξάρτητο μηχανισμό για το κράτο δικαίου στο μέλλον σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχουν κυρώσει για αυτού που δεν σέβονται τι βασικέ μα αρχέ. Αυτό είναι το πιστεύω μου. Ευχαριστώ, Μάνφρετ Βέμπερ. Γιάννη Ζαχράντιλ, εκ μέρου ε, των μεταρρυθμιστών συντηρητικών. Θέλετε να προσπιστείτε την Ευρώπη. Το κύριο πρόβλημα για μένα είναι ότι οι απλοί άνθρωποι, οι πολίτες της χώρας μας δεν ενδιαφέρονται για κάθε μέρα για την πολιτική αλλά τους έχει κουράσει η ατελείωτη ευρωπαϊκή ενοποίηση. Βλέπουν ότι παρεμβαίνει η Ευρώπη στην καθημερινότητά τους και απειλεί τις παραδόσεις τους, τα έθιμά τους. Βεβαίως είμαι λοιπόν υπέρ της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της ευρωπαϊκής ενότητας, αλλά όπως είπα από την αρχή, θέλω μια Ευρώπη να κάνει λιγότερα καλύτερα. Μια Ευρώπη που να είναι πιο αποκεντρωμένη, πιο ευέλικτη. Δεν είναι η καλύτερη απάντηση σε κάθε πρόβλημα περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη, όπως προτείνει το ΕΛ και οι σοσιαλιστές, που είναι αυτοί που τα τελευταία 25 χρόνια είναι υπεύθυνοι για την πορεία τη Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν τη στάση τους. Ευχαριστώ, Φραν Τίμερμανς. Παρακαλώ. Νομίζω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η διαφορά των απόψεων σε ό,τι αφορά την πολωνική κυβέρνηση ε, που υπήρχε τα τελευταία τρία χρόνια. Ο κόσμο έλεγε ότι αχ, μην τα κάνετε αυτά γιατί θα απογοητεύσετε τον κόσμο. Ο κύριο Ζαχραντέλη πώ εξηγεί όμω το γεγονό ότι μετά από τρία χρόνια πολύ σκληρών ε, διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση αυτή, η υποστήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολωνική κοινωνία είναι πολύ πιο υψηλή. Ο πολωνικό λαό μα δίνει πιο πολύ σημασία από πριν. Θέλουν να είναι τμήμα αυτή τη κοινότητα των αξιών. Να του το δώσετε αυτό, μην του το κρατάτε αυτό. Ε, Uh, Από πλευρά ε, των Πολωνών, να σα δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Από τη δική μου τη χώρα, 90% των Τσέχων πολιτών θέλουν προφανώ να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι του αρέσει η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση κατά κάποιο τρόπο, ενώ 75% των πολιτών τη Τσεχία δεν θέλουν να υιοθετήσουν το ευρώ. Είναι ένα σαφέ παράδειγμα ότι στον κόσμο του αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν του αρέσουν όλα όσα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο εθνικό επίπεδο. Και δυστυχώ αυτό έχει ανατραπεί υπέρ τη ευρωπαϊκού επίπεδου. Ευχαριστώ πολύ. Μαγκρέτε Βεστάγκερ. Τι έχει απομακρύνει του πολίτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι αυτοκριτική έχετε να κάνετε. Πολλοί είναι οι λόγοι νομίζω. Αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τον εαυτό μας τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε. Πολύ συχνά μιλάμε σαν να έχουμε κάτι κρυφό να κρατήσουμε μυστικό, με διάφορα κρονίμια. Να, πέρσι ξεκινήσαμε με τα ε, ψηφιακά δικαιώματα του πολίτη και δώσαμε τον τίτλο στον κανονισμό GDPR. Πώς θα το καταλάβει αυτό ο πολίτης. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο με τον οποίο μιλάμε, να βγάλουμε τις ετικέτες και τους τίτλους αυτούς. Ιδάλλως ο κόσμος θα πει, μα Πού είναι το πρόβλημα. Να, να το περιγράψουμε το πρόβλημα και να καταλάβει ο κόσμο τι είναι και να του πούμε την αλήθεια. Και να δείξουμε τι συμβαίνει, να καταπολεμήσουμε όλα αυτά τα ε, fake news, τα ψεύτικα νέα ή την παραπληροφόρηση που κυκλοφορεί, να δώσουμε ουσία στη συζήτηση, τροφή σκέψη στον πολίτη, να ξαναβάλουμε στο επίκεντρο το πώ θα ξαναγυρίσουμε στη δημοκρατία, πώ θα βελτιώσουμε τη δημοκρατία στην καθημερινή ζωή. Ευχαριστώ. Έχουμε καθυστερήσει πολύ γρήγορα στην Αναστήνα. Τι γίνεται στα κοινωνικά μέσα. Κοιτάξτε, έχουμε χιλιάδε ε, άτομα που μα στέλνουν μηνύματα. 5.000 άτομα παρακολουθούν το YouTube, 28.000 στο Facebook, 7.000 στο Twitter. Και ω τώρα να σα πω ότι έχουμε κορυφαίε θέσει στο Βέλγιο, στη Δανία, την Ιρλανδία, στην Φιλανδία, Κύπτος και πολλοί μας στείλατε ερωτήσει για συγκεκριμένα θέματα, αλλά και πολλοί μας ε, θέτετε διαφορετικά, πιο ευραία θέματα. Για παράδειγμα, από την Ιταλία έχουμε μία ερώτηση από έναν ε, πολίτη της Ευρώπης που μας λέει γιατί να θεωρώ ότι με εκπροσωπούν τα εθνικά σας κόμματα. Ευχαριστώ και σας δίνω το λόγο. Μια τελευταία ευκαιρία αγαπητοί υποψήφοι τώρα για να ζητήσετε την υποστήριξη του πολίτη για την επόμενη πενταετία στη θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής, Φραν Τίμερμανς. Ε, 40, 40 δεύτερα μόνο, γιατί το ένα λεπτό δεν μπορούμε να το διαθέσουμε, έχουμε καθυστερήσει. Μας ακούσατε σήμερα. Ακούσατε τις διαφορές μας. Ελπίζω να σας βοηθήσει να αποφασίσετε πώς θα ψηφίσετε την επόμενη εβδομάδα. Ένα πράγμα όμως θέλω να σας ζητήσω. Όποιον και να επιλέξετε, να μην γίνετε αδιάφοροι, να επιλέξετε, να ακουστεί η φωνή σας. Αν δεν ψηφίσετε, κάποιος άλλος θα μιλήσει για σας. Είναι σαν να δίνετε τα χρήματά σας σε κάποιον άλλον για να τα ξοδέψει. Ψηφίστε. Ψηφίστε από την καρδιά σας. Ψηφίστε για το κόμμα ή το άτομο που θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα. Αλλά ψηφίστε. Μην γίνετε απαθείς. Manfred Weber. Αν είχα την ευκαιρία να ρωτήσω τη γενιά των παππούδων μας τι σκέφτονται για την ε, τωρινή Ευρώπη, ξέρω ότι θα λέγανε είναι η καλύτερη Ευρώπη που είχαμε ποτέ. Και τώρα με τις εκλογές αυτές έχουμε την ευκαιρία να την υπερασπιστούμε κατά των εγωισμών, κατά των εθνικισμών και να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο. Θέλω να ανοίξω ένα κεφάλαιο με αισιοδοξία, με προοπτική για το μέλλον, για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτή την υπέροχη ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης και το είπα και πάλι. Θέλω αυτό να γίνει με τρόπο δημοκρατικό. Εσείς αποφασίζετε, εσείς θα αποφασίσετε και για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εσείς θα δώσετε την καθοδήγηση για τα κύρια θέματα που θα μας απασχολήσουν στο δημόσιο διάλογο στην επόμενη πενταετία. Μια πραγματικά γνήσια, δημοκρατική Ευρώπη και ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία Βεστάκερ. Δύο πράγματα. Καταρχά, είναι σημαντικό να δείξουμε ότι αλλάζουμε και ο πιο προφανή τρόπο να το κάνουμε είναι να έχουμε μια επιτροπή με ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Αυτό αποτυπώνει τις κοινωνίες μας και κατά δεύτερον αυτά που συζητάμε σήμερα, τα θέματα που συζητάμε σήμερα είναι δύσκολα θέματα. Χρειαζόμαστε να το κάνουμε. Αλλά χρειάζεται τόλμη, χρειάζεται θάρρο για να ξεπεράσουμε τον εαυτό μα και να ξεπεράσουμε και τι διαφορέ μα, να βρούμε κοινέ λύσει. Η δύναμη να αλλάξουμε είναι δική σας, από σας έρχεται. Το να ψηφίσει κανείς είναι δύναμη. Να ψηφίσετε λοιπόν στις εκλογές αυτές και να εμπνεύσετε και άλλο κόσμο να ψηφίσουν. Γιατί άλλο, ε, άλλοι θα το χρησιμοποιήσουν άλλοι το δικαίωμα αυτό. Ευχαριστώ. Ίσως ε, κανείς από τους παρόντες εδώ δεν ε, είναι ικανοποιημένος από το πώς είναι τα πράγματα στην Ένωση. Αλλά ο καθένας μας έχει άλλη συνταγή για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η χώρα μου εντάχθηκε στην Ένωση πριν από 15 χρόνια. Είμαι από άλλο τμήμα της Ευρώπης. Με διαφορετικές εμπειρίες και με διαφορετικό τρόπο αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ίσως ε, δεν είναι ευρέω κατανοητό αυτό σε άλλα τμήματα της Ευρώπης ότι είμαστε πιο ευαίσθητοι για θέματα κυριαρχία και εθνικής ταυτότητας για να συνεργαστούμε και για να ζήσουμε μαζί πρέπει να βρούμε τρόπο για να έχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επίπεδου, όπως είπα και στην αρχή. Ευχαριστώ πολύ, Σχακέλε. Παντού στην Ευρώπη οι νέοι βγαίνουν στους δρόμους γιατί φοβούνται, φοβούνται και το μέλλον τους. Και στρέφουν αυτό το θυμό προς τους πολιτικούς που δεν κάνουν κάτι. Θέλουν λοιπόν να μετατρέψουν το θυμό αυτό σε δράση. Και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς, να δράσουμε, γιατί υπάρχει ελπίδα για καλύτερο μέλλον και μπορούμε να το πετύχουμε. Αλλά χρειάζεται αλλαγή και χρειάζεται θάρρος. Και χρειάζεται και μια ισχυρή φωνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα αγωνιστεί για την προστασία του κλίματο για την κοινωνική Ευρώπη, και για τη δημοκρατία. Όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Και αυτό είναι που έχουμε να προσφέρουμε ως πράσινη προς όλους τους Ευρωπαίους. Ο Νίκο μόλις τι συμβαίνει. Οι ηγέτε, οι Ευρωπαίοι μιλούν, αλλά δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα. Την κλιματική αλλαγή, τι επισφαλεί θέσει εργασία, τη φοροαπάτη και φοροδιαφυγή. Εμεί θέλουμε μια Ευρώπη που θα δίνει απαντήσει σε όλε αυτέ τι προκλήσει. Θέλουμε στην Ισπανία να δοθεί ψήφο για την Ευρώπη, για το φεμινισμό. Στην Ιταλία να δοθεί ψήφο για την Ευρώπη και για αντίσταση στο φασισμό. Θέλουμε σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη να δοθεί ψήφο για το κοινωνικό κράτο που θα, τους, θα επιτρέψει τους πολίτες να ζουν με αξιοπρέπεια. Θέλουμε να αλλάξει ρότα η Ευρώπη. Θέλουμε ε, ψήφο για την Ευρωπαϊκή Αριστερά που είναι η μόνη η οποία μπορεί να αλλάξει τη ρότα της Ευρώπης. Ευχαριστώ Νίκο Κουέ. Έληξε η συζήτησή μα. Ελπίζω να σα βοήθησε να κάνετε την επιλογή σα για τον επόμενο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτηση. Αλλά, εν πάση σα παρακαλώ να δείξουμε όλη την εκτίμησή μα προ όλου του έξι υποψηφίου. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την συζήτηση, το debate. Για να δούμε, Αναστήνα, τι έγινε στο διαδικτύο. Ήταν πολύ ζωή η συζήτηση. Δεν μπορέσαμε να τα σημειώσουμε όλα, αλλά πολλοί από εσά ζήτησαν μεγαλύτερη κάλυψη για τι ευρωεκλογέ. Και επίση, τρει ε, από δημοσιογράφου από τη Γαλλία και τη Γερμανία ανέφεραν ότι η σημερινή συζήτηση αποτελεί μια συζήτηση σεβασμού γεμάτη νόημα. Ευχαριστούμε. Και σε όλους σας εδώ, στο Κοινοβούλιο, αλλά και σε, εμάς που, σε που παρακολουθείτε από το σπίτι, ψηφίστε 23 με 26 Μαΐου, ανάλογα με τη χώρα σας. Και από την ομάδα της Eurovision για το ευρωπαϊκό debate, καλή σας νύχτα. Bonsoir, good night.